Καλημέρα συνάδελφοι. Πολύ διαφορετικά φαίνεται η αίθουσα από το Προεδρείο, από το έδρανο, από, ότι, από χαμηλά, από την αίθουσα. Και καλό είναι για την ΚΟΕ να προεδρεύσει καμιά φορά. Θα ζητήσω λοιπόν από τον Αντρέα Σφα που εκπροσωπεί τον εισηγητή να μας παρουσιάσει το θέμα. Καλημέρα συνάδελφοι, χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαστε εδώ στην ίδια σύνθεση όπως εχθές το βράδυ, απλώς σε διαφορετική αίθουσα. Γι' αυτό θα ε, προσπαθήσω να σας παρουσιάσω το θέμα των ενεργειακών αγορών, διαφάνεια και επάρκεια στα αγγλικά. Για να μην έχουμε, έχετε ανάγκη των ακουστικών σας. Θα ήθελα λοιπόν καταρχάς να πω ότι αυτός ο κανονισμός προσπαθεί να δημιουργήσει ένα πλαίσιο και να αποφύγει την κατάχρηση των αγορών όπως ας πούμε τις ε, παράνομες εσωτερικές ε, συναλλαγές, ε, την απόκρυψη θεμητών συναλλαγών και άλλα, άλλες παραβάσεις. Αυτές οι αγορές ε, επηρεάζουν... Α, ε, τώρα, ε, ναι, στα γερμανικά. Θα μιλήσω λίγο αργότερα. Αυτές οι αγορές οπωσδήποτε επηρεάζουν την ευημερία των πολιτών και την ποιότητα ζωής τους, δεδομένου ότι άπτονται της ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού αερίου κλπ. Άρα λοιπόν πρέπει να αποφύγουμε πάση θυσία κατά χρήση της αγοράς αυτής και να εξασφαλίσουμε την ακεραιότητα και την αξιοπιστία. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία των αγορών ενέργειας και να εγγυηθούμε θεμητές τιμές τους χρήστες, τους καταναλωτές. Τα μέτρα λοιπόν που προτείνονται εδώ είναι καταρχάς εποπτεία της αγοράς για να διαπιστώσουμε αν υπάρχει κατάχρηση πρέπει καταρχάς να έχουμε ένα σωστό σύστημα εποπτείας ε, διασυνοριακών συναλλαγών και ε, δεδομένων για να κατανοήσουμε απόλυτα τις ε, εξελίξεις που γίνονται σε αυτή την αγορά η αρχή, η ΕΣΑ πρέπει να έχει πρόσβαση σε όλες τις διμερείς συμφωνίες και ιδίω στο άρθρο 14 της συνθήκης το οποίο, ε, του κανονισμού συγγνώμη, το οποίο προβλέπει κυρώσεις. Κυρώσεις στην περίπτωση παραβάσεων και καταχρήσεων οι οποίες ε, κυρώσεις πρέπει να είναι ανάλογες της παράβασης. Η στον υπολογισμό αυτών των κυρώσεων πρέπει να ληφθεί υπόψη και το μέγεθος της ζημίας προς τους καταναλωτές. Λοιπόν, εποπτεία κυρώσεις και το τρίτο σημείο στο οποίο επικεντρώνεται η έκθεση είναι η Κομισιόν. Η οποία μπορεί να αναθέσει, ε, να, να προτείνει νομοθετικές ε, πράξεις, ε, την συλλογή δεδομένων, και ο κανονισμός επιτρέπει στην Κομισιόν να υιοθετήσει αυτές τις πράξεις. Πρόσφατα έχει υπογραφεί το μνημόνιο της, ε, που δίνει τη δυνατότητα υπογραφής ε, ε, πράξεων και εάν υπάρχουν εφόσον η Κομισιόν συνυπογράψει ε, αυτές τις ε, πράξεις, πρέπει να φροντίσει και για την ε, μεταφορά τους στους ενδιαφερόμενους και την υποβολή τους στις ενδιαφερόμενες υπηρεσίε. Αυτά λοιπόν είχα να σας πω μετά από την παράκληση του εισηγητή να τον αντικαταστήσω. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ και ε, από τώρα προχωράμε στους κοιόδης εισηγητές, ο κύριος Παντσέρη από τους Σοσιαλιστές. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή και μέσω του εκπροσώπου του ακριβώς για να τον ευχαριστήσει με τη σειρά του για την ε, όρεξή του, την όρεξη που έδειξε, τη διάθεσή του και επίσης με τους κοινοσυγητές στο Στρασβούργο μας έδωσε πολύτιμες ενδείξεις και όσα είπαμε νομίζω βλέπω ότι έχουν περιληφθεί ήδη στην έκθεσή του. Όλα αυτά είναι θετικά γιατί αυτό που κάνουμε εμείς ε, αφορά την προστασία των καταναλωτών δηλαδή περισσότερη διαφάνεια και σωστό χαρακτήρα της αγοράς ε, από τη στιγμή που δεν θα γίνουν σεβαστά ορισμένα πράγματα τότε θα υπάρξει μια αποζημίωση όσον μετά από την ζημιά που θα υποστούν οι καταναλωτές στο άρθρο 2 και αυτό είναι σημαντικό αναφέρονται πράγματα σημαντικά και θα πρέπει να υπάρξει μια μεταβίβαση των ε, ε, στοιχείων στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο για να υπάρξουν διάφανες διαβουλεύσεις. Συνολικά έχει μπει στο σωστό δρόμο αυτή η έκθεση. Έχουμε ακόμα δύο σημεία που θα πρέπει να εκτιμήσουμε και που πιστεύω ότι χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες για να δούμε πώς αυτά τα δύο σημεία θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στην έκθεση. Ίσως θα χρειαζόταν να δείξουμε ότι αυτές οι κυρώσεις ουσιαστικά θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν ε, σε όλα τα κράτη-μέλη και όχι να κάνει κανείς διατησία ανάλογα, δηλαδή ανάλογα ε, να διαλέγει κανείς τη χώρα που θα κλείσει αυτές τις συμφωνίες επειδή θα υποστεί ενδεχόμενα τις ε, ελαφρότερες κυρώσεις γιατί έτσι θα στρεβλωθούν και οι κανόνες της αγοράς. Εδώ λοιπόν, ε, τελευταίο σημείο, πιστεύω επίσης ότι θα πρέπει να δούμε και τις μικροεπιχειρήσεις που διαφορετικά από τις μεγάλες επιχειρήσεις δεν μπορούν να διαπραγματευτούν τόσο ισχυρά με τους απέναντι και θα μπορούσαμε να έχουμε τις τροπολογίες 1 και 2, να κάνουμε μια συγκεκριμένη αναφορά ακριβώς στις μικροεπιχειρήσεις γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει και αυτή η αγορά που θα πρέπει οπωσδήποτε να προστατευθεί. Αυτά υπόλοιπα, ναι, κρινοθετική την έκθεση. Σας ευχαριστώ. Thank you, Mr. Σας ευχαριστώ κύριε Παντσέρη. Για την Άλτα. Δεν υπάρχει κανείς παρόν. Αυτή τη στιγμή προχωρούμε στους πράσινους. Α, τους Ευρωπαίους συντηρητικούς, και κ. Σάσλι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σφάμπ για την εισήγησή του και να ευχαριστήσει επίσης τον εισηγητή για το σχέδιο γνωμοδότησης. Είμαι... Είμαστε πολύ ευτυχείς που λαμβάνει υπόψη την προστασία των καταναλωτών αυτή η πρόταση και περιμένουμε και την γνωμοδότηση της ΙΤΡΕ. Θέλουμε οπωσδήποτε η αγορά να λειτουργεί σε ένα δίκαιο επίπεδο, διότι γίνονται πολλές διασυνοριακές συναλλαγές και διαπραγματεύσεις ε, ενεργειακών ανταλλαγών. Άρα λοιπόν άπτεται μιας κανονιστικής και μη κανονιστικής αγοράς. Ε, ε, εκτός οργανωμένων συναλλαγών γίνονται άλλες ε, συναλλαγές ευρύτατες. Άρα λοιπόν χρειάζεται ρύθμιση και ο, ο τομέας που δεν εμπίπτει στο κανονιστικό πλαίσιο και πρέπει να εξετάσουμε, να εποπτεύσουμε ε, εις βάθος ε, όλες τις δραστηριότητες αυτές ε, στο έδαφος της κοινότητας, της Ένωσης, έτσι ώστε οι καταναλωτές να πιστεύουν, να έχουν πίστη και να εμπιστεύονται την αγορά και να ε, υποφελούνται από δίκαιες και θεμητές τιμές. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ιδίω ε, σε περίπτωση κυρώσεων να λυθούν υπόψη σοβαρά οι τυχόν επιπτώσεις στους καταναλωτές. Τροπολογία 8. Ο εισηγητής έχει διαγράψει ε, ένα μέρος του κειμένου που πρότεινε η Επιτροπή αρχικά, όπου αναφέρονται οι σεμιτές πρακτικές, οι αποδεκτές πρακτικές στην οικία, ενεργειακή αγορά κλπ. Εντολές διαπραγμάτευσης συνάδουν με τις αποδεκτές πρακτικές. Πρέπει να το μελετήσουμε αυτό, διότι κατά εμέ το κλειδί είναι η διαφάνεια και με όσο, όσο αυξάνεται και βελτιώνεται η διαφάνεια, δεν νομίζω ότι κάποιος θα μπορεί να εφαρμόσει μη αποδεκτές πρακτικές. Αυτή ήταν η επιφύλαξή μου στην τροπολογία 8. Κατά τα άλλα συγχαίρω τον εισηγητή για, το, για την εργασία του. Α, ευχαριστούμε τον κύριο Φόξ. Ο επόμενο εισηγητή είναι ο κύριο Τριανταφυλλίδη ε, από την ΚΟΥ, εγώ δηλαδή, και από πρόοδο αλλάζω καπέλο και γίνομαι σκιώδη εισηγητή. Και μιλώ ελληνικά. Διαφάνεια στην ενεργειακή αγορά περιέχει μια σειρά από πολύ σημαντικές διαπιστώσεις. Το κεντρικό στοιχείο ανάλυσης είναι η διαπίστωση ότι αν και η μεταφορά της παραγωγής και εμπορίας ενέργειας διαμέσου των δευτερευουσών χρηματιστηριακών αγορών, ειδικά διαμορφωμένων μόνο για τον τομέα της ενέργειας, είχε θετικά αποτελέσματα, την ίδια στιγμή το εφιστάμενο καθεστώς έχει επιφέρει ελλείψεις στους εφαρμοστέους κανόνες και στο επίπεδο διαφάνειας. Πάγια μας θέση είναι η παροχή υψηλής ποιότητας ενέργειας σε προσιτές τιμές για τους πολίτες. Έχοντας ως αφετηρία το πιο πάνω, θα πρέπει να μας απασχολήσει το πώς η φύση τέτοιων αγορών συνάδει με το πιο πάνω στόχο και κατά πόσο είναι εφικτή η επίτευξη προσιτών τιμών για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν αυτές εξαρτώνται από κερδοσκοπικές πιέσεις σε αυτές τις αγορές. Παράλληλα αποδεικνύεται η ύπαρξη αδιαφάνειας μέχρι και σχρογκέρδειας η οποία διονγκώνεται μέσα από τις χρηματιστηριακές πράξεις. Άρα είναι αναγκαία η θέσπιση μέτρων που να αντιστρέφουν την κατάχρηση και όχι απλά να την ρυθμίζουν. Η ενίσχυση των χρηματαγορών στον ενεργειακό τομέα θα αυξάνει και τους κινδύνους που παρουσιάζουν τέτοιες αγορές. Συνεπώς η δράση μας θα πρέπει να επικεντρωθεί σε ιδιαίτερα μέτρα για την προστασία των καταναλωτών, ενισχύοντας τη διαφάνεια και εξελίσσοντας την αποδοτικότητα της αγοράς. Τούτο σημαίνει χαμηλότερο κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Θα πρέπει όμως να έχουμε πάντοτε κατά νου τη διαφορετικότητα στην οργάνωση των αγορών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κλείνοντας, θα ήθελα να κάνω ιδιαίτερη αναφορά στις κυρώσεις για χειραγώγηση της αγοράς. Θα πρέπει να υπάρξει μια ευθυγράμμιση, έχοντας όμως κατά νου ότι ο ενεργειακός τομέας συμπεριλαμβάνει ισχυρές εθνικές ρυθμιστικές αρχές, όπου ήδη είναι επιφορτισμένες με αυτό το ρόλο. Μια ρύθμιση που θα καταργεί το ρόλο που διαδραματίζουν οι εν λόγω αρχές σήμερα θα αποτελέσει πίσω γύρισμα στις προσπάθειες για εποπτεία και διαφάνεια στις ενεργειακές αγορές. Now Mr. puts on his hat και τώρα ξαναφοράω το καπέλο του Προέδρου και βλέπω ότι ήρθε ο κύριος Τούμες από τους πράσινους και του ζητώ να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, συγχαίρω τον κύριο Σκόφσκι για τη γνωμοδότησή του. Νομίζω ότι είναι πολύ καλά συντεταγμένη και ως ΙΜΚΟ πρέπει να την προσέξουμε. ιδίω. Ιδίως για τα μη δομημένα προϊόντα, τα αυτά τα οποία δεν εμπίπτουν στο κανονιστικό πλαίσιο, υπάρχουν πολλές ε, συναλλαγές εκτός κανονιστικού πλαισίου και εντός βεβαίως, οπότε πρέπει να αυξήσουμε τον έλεγχο για να ξέρουμε ότι τα απαραίτητα δεδομένα τα στέλνονται στην Ευρωπαϊκή Αρχή, ε, αρμόδια αρχή προς εξέταση. Επίσης, η προστασία των καταναλωτών ε, πρέπει να ληφθεί υπόψη στην επεξεργασία των κυρώσεων, διότι γίνεται χειραγώγηση των αγορών και εκατομμύρια, εκατομμύρια ευρώ ε, αρπάζονται από τις τσέπες των καταναλωτών με αυτές τις ασέμητες συναλλαγές. Πρέπει λοιπόν να λάβουμε σοβαρά υπόψη τις επιπτώσεις στους καταναλωτές. Πολύ σημαντικά ε, στοιχεία αυτά, τα δύο, στην ε, γνωμοδότηση. Τα περισσότερα σημεία της έξεσης ε, συμφωνούμε, μία-δύο τροπολογίες ίσως θα υποβάλουμε, τροπολογία 18 εδώ γίνεται μία διασύνδεση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Αρχής, ε, την ΕΣΜΑ και της ΕΣΑ και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών και της ΕΣΑ ε, πρέπει να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να ρυθμίσουμε τα θέματα αυτά ε, και μέσω των χρηματοοικονομικών αγορών. Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι δεν χρειάζεται η, να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Αρχή Αξιών και Αγορών, αλλά ιδίω για τους μεγάλους οργανισμούς, τους μεγάλους εμπορευόμενους των αγορών αυτών, ε, μην ξεχνάμε ότι επενδύουν σε παράγωγα ε, προϊόντα, χρηματοοικονομικά προϊόντα, σε προθεσμιακά προϊόντα. Άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε το μάτι μας και σε αυτά, σε αυτή την αγορά ε, πολλές φορές αυτές, αυτοί οι οργανισμοί ε, δεν θέλουν ή δημιουργούν προβλήματα στην υποβολή των στοιχείων τους ε, στην ESA, στην Ευρωπαϊκή Αρχή. Ε, δεν νομίζω λοιπόν ότι η συμπερίληψη της ΕΣΜΑ δημιουργεί παραπάνω γραφειοκρατία, επιπλέον γραφειοκρατία. Πιστεύω ότι χρειάζεται όλες αυτές οι ανταλλαγές πληροφοριών χρειάζονται ε, και από τις ρυθμιστικές αρχές και από τις αρμόδιες οικονομικές αρχές των κρατών μελών. Γενικά ευχαριστώ τον εισηγητή και τον συγχαίρω για τη γνωμοδότησή του. Ευχαριστώ κύριο Τούμες. Κανένας άλλος δεν ζήτησε το λόγο και δίνω το λόγο στον εκπρόσωπο της Κομισιόν, τον κύριο Ομπράιεν νομίζω. Uh, uh, Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την έκθεση και για την υποδοχή των προτάσεών μας. Με μεγάλη χαρά διαπιστώσαμε τα σημεία που θέσατε στην έκθεσή σας. Πολλά από αυτά έχουν ήδη συζητηθεί με τα κράτη-μέλη και με τους ε, συναδέλφους σας της Επιτροπής Ήτρα. Εδώ Αναφερθήκατε συγκεκριμένα και θεωρήσατε ότι είναι ευπρόσδεκτη η ACERS ή ο οργανισμός για, τη για... που θα ασχολείται με τα στοιχεία των συναλλαγών. Είναι χρήσιμο για να μπορεί να επιβλέπει μια εκτεταμένη σειρά συναλλαγών και στοιχείων συμπεριλαμβανομένων και των συναλλαγών OTC. Ε, τώρα, όσον αφορά τις διατάξεις, πράγματι οι ομάδες εργασίες εργάστηκαν και εντόπισαν την ανάγκη για περαιτέρω ε, εναρμόνιση στις διατάξεις που αφορούν τις ποινές. Είχαμε και τη συνεργασία των συναδέλφων της Γενικής Διεύθυνσης Market που μελέτησαν ε, στο πλαίσιο της πρόσφατης αναθεώρησης του χρηματοοικονομικού κανονισμού. Πήραμε στοιχεία και από εκεί. Έχουν προχωρήσει. Αν μελετήσετε προσεκτικά το κείμενό μας γίνεται ε, συγκεκριμένη αναφορά στην αιτιολογική σκέψη 23 ε, στο ότι τα κράτη-μέλη που έχουν διατάξεις που αφορούν ποινές θα ευθυγραμμίζονται με αυτές του χρηματοοικονομικού κανονισμού γίνεται μια αξιολόγηση της ζημιάς εδώ στα πλαίσια, σε, σε, σχέση και με αυτό που υφίσταται το καταναλωτής. Αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα ιδέα. Επίσης, σκοπός μας είναι να επιμείνουμε ε, στην συνεννόηση που έγινε μεταξύ των θεσμικών οργάνων και έτσι το κείμενο παραμένει συνολικά συμπεριλαμβανομένων και των ιδεολογικών σκέψεων. Άρα, για μία ακόμα φορά σας ευχαριστώ πολύ για τη δουλειά σας και τις ενδιαφέρουσες προτάσεις σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Χούπερ. Τώρα θα, δώσω, θα ζητήσω στον εκπρόσωπο του ε, εισηγητή, τον κύριο Σβάπ, να, το λόγο για να κλείσει τη συζήτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη θετική αντιμετώπιση σας ε, εδώ στην αγορά αυτή στην Ευρώπη δεν είμαστε στο σημείο που θα θέλαμε. Γι' αυτό ακριβώς οι προτάσεις της Επιτροπής ε, που από τον εισηγήματα κρίνονται θετικές είναι κάτι το καλό. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε ώστε η ενέργεια ότι ώστε αυτό το κείμενο να γίνει δεκτό από όλη την Ευρώπη ακριβώς και να είναι μια σωστή ε, τοποθέτηση. Εδώ ε, το ξέρουν οι φυσικιώτες ηγητές πότε θα γίνει αυτό. Ε, λοιπόν, το μόνο που μένει να κάνω είναι να δηλώσω ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι 19η Απριλίου και να παραδώσω στον κύριο Μάλκον Χάρπερ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τον Κυριάκο για το γεγονός ότι προείδρευσε. Λοιπόν, ο κύριος Κρότσμαν, ο οποίος δεν είναι εδώ. Κύριε Τόρνες, είναι έτοιμη να φύγει. Πρέπει να δούμε πού είναι ο κύριος Κρότσμαν. Α, νάτος. Πάνω στην ώρα. Just let Λοιπόν, να αφήσουμε τον κύριο Κρότσμαν να κάτσει και μετά να παραλάβουμε το θέμα του. Good. Let's now move on to... Οπότε περνάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Έχουμε μεγάλη ποικιλία θεμάτων σήμερα το πρωί. Πρόκειται για μια γνωμοδότηση ε, για τον Ευρωπαϊκό Κινηματογράφο στην ψηφιακή εποχή. Ο μέγας ε, κινηματογραφόφιλός μας είναι ο κύριος Κρότσμαν, ο οποίος ε, είναι συντάκτης της Επιτροπής. Έχουμε τους Σκιώδης, Τουν, Βάιλερ, Ήσασταν εδώ χτες. Σας έψαχνα. Η κυρία Μακλάκιντ, Fox, καλύπτει τα θέματα του κινηματογράφου. Πολύ ωραία. Σαβίνη. Η κυρία Ρούλο δεν είναι εδώ. Η οποία έχει νομίζω τον τίτλο της σκιώδους εισηγήτριας της, της χρονιάς. πάση περιπτώσει, ο κύριος Κρότσμαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαστε, άργησα γιατί είναι εδώ μια αντιπροσωπή από την Ινδία και μιλούσα μαζί τους. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Θα συνεχίσω μιλώντας γερμανικά ε, για το θέμα τη ψηφιοποίηση του Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου. Εδώ στην εργασία μου αυτό που τονίζω είναι ότι ο κινηματογράφος δημιουργεί καινοτομία, δημιουργεί θέσεις εργασίας καινούριε. Αυτή η ψηφιοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο προωθεί δραστηριότητες ιδιαίτερα σημαντικές πολιτιστικές. Ταυτόχρονα αυτή η ψηφιοποίηση βοηθάει τον, την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού κινηματογράφου Ταυτόχρονα βέβαια ναι, αυτή η μορφή δεν θα πρέπει να θίγει άλλες μορφές. Αυτό που τονίζουμε είναι ότι θα πρέπει να λαμβάνουμε πάντα μέτρα υπέρ της αλλαγής στην ψηφιοποίηση και να επικεντρώσουμε την προσοχή μας ακριβώς στον κινηματογράφο αυτό καθ' αυτό. Να δούμε όταν δεν μπορούμε να έχουμε ενακτικές πηγές χρηματοδότησης εδώ το πέρασμα ψηφιακό θα πρέπει να γίνει όσο γίνεται συντομότερα και το κόστος θα πρέπει να κρατηθεί χαμηλό. Και τα κράτη-μέλη σε περίπτωση που το κράτος θα βοηθήσει να, προσέξουν τον ανταγωνισμό για να αποφύγουμε στρεβλώσεις της αγοράς και η Επιτροπή στη συνέχεια θα πρέπει να δείξει Ποιε είναι οι καθαρέ κατευθύνσει από νομική πλευράς. Δεν θα πρέπει όμως να έχουμε παρεμβάσεις στα κράτη-μέλη. Η προώθηση αυτής της ψηφιοποίησης πως απαιτεί η τεχνολογία να είναι κάτι το ουδέτερο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό δεν θα πρέπει να υπάρχουν ε, φόρμα που να ε, προτιμώνται από άλλα. Ταυτόχρονα χρειάζεται να συνεχίζονται οι χρηματοδοτήσεις, ε, να δούμε ακριβώς ποια είναι τα ειδικά χαρακτηριστικά στις αίθουσες προβολής και στους διανομής. Επίσης θα πρέπει να προσέξουμε σε διεθνώς επίπεδο και να αναπτύξουμε τα πρότυπα που να είναι συμβιβάζονται ακριβώς να μπορούν να συνδυαστούν με τις δυνατότητες προβολής. Υπάρχουν ε, standard ISO και η χρησιμοποίηση αυτή αυτόν το στάνταρτ στην ευρωπαϊκό κινηματογράφο θα μπορούσε να προωθηθεί. Εδώ Πρόκειται για πληροφορίες ε, που μου λένε ταυτόχρονα ότι υπάρχουν μονοπόλια των διανομέων που έχουν αναπτύξει αυτά τα πρότυπα για την ψηφιοποίηση. Ίσως ακριβώς είναι αυτά τα μονοπόλια που κυριαρχούν στην αγορά. Εάν υπάρχουν προδιαγραφές που όλοι να δέχονται, τότε μπορούμε να αναφερθούμε σε αυτές για να αποφύγουμε τα εμπόδια στις προτάσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κρότσμαν. κύριε Τούν. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ για την προσφορά του κυρίου Κρότσμαν. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα. Και εν μέρη πρέπει να παραδεχτώ ότι εμπλέκομαι προσωπικά, γιατί στη δική μου εκλογική περιφέρεια υπάρχει ένα πολύ πυκνό δίκτυο ψηφιακών κινηματογράφων που μοιάζει ότι να έχει αλλάξει τη ζωή πολλών κατοίκων, ιδίω των απομακρυσμένων περιοχών. Πέρυσι το Σεπτέμβριο οργάνωσα εδώ μια διάσκεψη για το ψηφιακό μέλλον του ευρωπαϊκού κινηματογράφου και καταλήξαμε σε πολλά χρήσιμα συμπεράσματα, πολλά από τα οποία συμπεριλάβατε και εσείς στην ε, γνωμοδότησή σας. Θα ήθελα όμως να υπογραμμίσω, επειδή είμαι και μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού, ε, υπάρχει λοιπόν και αυτή η πολιστική διάσταση την οποία θέλω να υπογραμμίσω λίγο περισσότερο ε, σε σχέση με τον ψηφιακό κινηματογράφο. Η, μεγάλη, πολύ μεγαλύτερη προ, εύκολη πρόσβαση και φθηνότερη ε, ε, πρόσβαση στον κινηματογράφο. Η, το γεγονός ότι μεγάλα πολιτιστικά ε, μεγάλες πολιτικές εκδηλώσεις όπως όπερες μπορούν να μεταδοθούν ε, σε πραγματικό χρόνο σε απομακρυσμένες περιοχές. Επίσης τα, οι αγώνες ποδοσφαίρου ή την Πρωτομαγιά ε, όταν θα γίνει τελετή με τον Πάπα. Υπάρχει κόσμος που έχει πρόσβαση σε πολύ μακρινά γεγονότα στα οποία ονειρεύεται ότι μπορεί να παρευρεθεί. Υπάρχει λοιπόν ένα πολιτιστικό σκέλος αυτή την όλη ιστορία. Οι μικροί αυτοί κινηματογράφοι ε, γίνονται χώροι ε, συγκέντρωσης ανθρώπων σε περιοχές όπου δεν συμβαίνουν πολλά πράγματα. Πρέπει λοιπόν ε, να υπάρξει ένα πλαίσιο οικονομικής και χρηματοδοτικής στήριξής τους. Αυτό πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο. Κάτι άλλο που θέλω να προσθέσω στη δική σας γνωμοδότηση είναι ότι όλοι γνωρίζουμε το πρόγραμμα Media. Η Κομισιόν αυτή τη στιγμή συντάσσει ένα νέο πρόγραμμα Media για το 2014. Πολλοί από εμά θα έχουμε ακούσει ότι ο κόσμος του κινηματογράφου ανησυχεί επειδή υπάρχουν φήμες περιορισμού μείωσης του προγράμματος. Εγώ ε, λέω μήπως να το βάλουμε ε, να το συμπεριλάβουμε στη γνωμοδότησή μας, ότι στηρίζουμε την περαιτέρω χρηματοδότηση του προγράμματος Media, διότι αυτό πραγματικά ενισχύει την ανάπτυξη ε, αυτού του τύπου, δηλαδή στηρίζονται οι μικροί κινηματογράφοι, οι παραγωγές, η ε, διακίνηση κλπ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Um, ευχαριστώ. Δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσο, ότι έχουμε τόσο σπουδαίους ειδικού εδώ. Η κυρία Βάιλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν είμαι ιδιαίτερα έμπειρη, αλλά καταναλώνω πολύ κινηματογραφό και η έκθεση του κυρίου Κρόιτσμαν αποτελεί μια πολύ καλή βάση για τη συζήτησή μας. Θα ήθελα να προσφέρω ορισμένα άλλα στοιχεία συμπληρωματικά. Θα πρέπει στην Επιτροπή μας να λάβουμε υπόψη μας ε, θέματα τα οποία, με τα οποία ασχολείται η Επιτροπή Πολιτισμού, πολιτιστικών θεμάτων, αλλά δεν θα πρέπει να ε, παραγνωρίζουμε και τα θέματα τα κοινωνικά για την βιομηχανία του κινηματογράφου ακριβώς. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες καινοτομία, ανάπτυξης κλπ. Το καταλαβαίνω αυτό, αλλά δεν πρόκειται μόνο για αυτό το θέμα. Αλλά όχι μόνο σε ε, γεωγραφικές ε, περιοχές οι οποίες διατρέχουν κίνδυνο. Είναι ασαφής αυτός ο ορισμός. Τι εννοούμε με αυτόν τον ορισμό. Εννοούμε την Ήπεθρο, έτσι αλλά όχι μόνο στην Ήπεθρο, στις ε, απομακρυσμένες περιοχές πεθαίνουν οι κινηματογραφικές αίθουσες, αλλά και στις μεγάλες πόλεις, στα αστικά κέντρα. Υπάρχουν κινηματογραφικές αίθουσες που δεν μπορούν να προσαρμοστούν στην ψηφιακή εποχή. Και πρέπει να προσέξουμε και τα μικρά σινεμά, τα τέχνης, τα οποία ε, με τα βίας επιβιώνουν και πρέπει να προβάλλουν ευρωπαϊκά έργα. διότι ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος είναι ένα σπουδαίο ανταγωνιστικό εργαλείο έναντι του, της Αμερικής και της Ασίας και των δικών τους παραγωγών. Θέλουμε λοιπόν να βοηθήσουμε και να ενισχύσουμε τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο. Εν συνεχεία κύριε Κρότσμα, στο σημείο 3 λέτε ότι θα πρέπει η μεταβατική περίοδος να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη σε σχέση με τις ε, ευαίσθητες ή υπαίθριες ας πούμε περιοχές και εν συνεχεία δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το ΕΦΡ. Υπάρχουν, υπάρχει το διαθροτικό ταμείο, το ΕΦΡ ήταν ένας βασικός μοχλός ε, στήριξης αδύναμων ε, ε, κινηματογραφικών αιθουσών ή αλυσίδων. Τέλος πάντων πρέπει να προβάλλουμε ε, την μεγάλη ε, επιτυχία της ΕΦΡΕΜ. Επίσης ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να ρυθμίσουμε το θέμα των προτύπων. Οπωσδήποτε αυτό είναι σημαντικό για τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο. Να μην, να μην λειτουργούν οι τρεις μεγάλες κινηματογραφικές περιοχές με διαφορετικά πρότυπα. Χρήση λοιπόν ενιαίων προτύπων. Πιστεύω ότι η έκθεση αυτή θα είναι ουσιαστική και θα συμβάλλει στην επιτυχία του ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Now, um... Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριος Φόξ. Θέλετε μήπως να πάρετε το λόγο εκ μέρους της κυρίας Μακλάρκεν. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, εκ μέρους της κυρίας Μακλάρκεν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κρόιτσμαν για την γνωμοδότηση αυτή που συνέταξε. Κυρίως η έμφαση έχει δοθεί σε σημείο διαφορετικό από ό,τι είχε δώσει η κυρία Βάιλερ. Εκείνη αναφέρθηκε στο κοινωνικό, πολιτιστικό ε, σκέλος. Αυτό είναι το, η δουλειά της Επιτροπής της. Εμείς πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα των καταναλωτών και της προστασίας των καταναλωτών. Γιατί καμιά φορά υπάρχει ο κίνδυνος όταν κάτι είναι πολύτιμο πολιτιστικά να υπάρχει η τάση να το επιδοτούν οι κυβερνήσεις. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι οι καταναλωτές είναι και φορολογούμενοι γιατί και είμαι ευγνώμων για την παράγραφο 4 της χρωμοδότησης του κυρίου Κρότσμαν. Πρέπει σαφώς να πούμε ότι βεβαίως υπάρχει το θέμα της επιδότησης των ε, ταινιών κλπ. Αλλά μένει αυτό στα κράτη-μέλη. ρόλο Κομισιών πρέπει να είναι να συντάσσει κατευθυντήριε γραμμέ που προτείνει ο κύριο Κρότσμαν. Όσο λιγότερα κάνει στον χώρο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο το καλύτερο. Πρέπει να εξασφαλίσουμε μια αγορά τεχνολογικά ουδέτερη, με τι λιγότερε δυνατέ επιδοτήσει και να μείνουμε εν αναμονή. Χαιρετίζω λοιπόν το έργο του κυρίου Κρότσμαν, κυρίω δε την παράγραφο 4 τη νομοθεσή του. Thank you very much. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα, ο κύριος Τριανταφυλλίδης, θέλετε το λόγο? Okay. Anyone else want to... Uh, uh, Mrs. Turner, did Mrs. Toon want to come back, yes? Yeah, of course. Yeah. Um, I'm sorry, but in the. Εγώ δεν θα έκανα στον τομέα αυτό τόσο αυστηρό διαχωρισμό μεταξύ του πολιτιστικού και του, ε, και της οικονομίας. Εσείς ε, στις, αυτές τις περιοχές που κινδυνεύουν εννοείται τις απομακρυσμένες, τις περιοχές της υπαίθρου. Αλλά επίσης όταν δεν συμβαίνουν πολλά πράγματα δεν αναπτύσσεται και η οικονομία. Αν η αν δεν κινητοποιείται, αν δεν δραστηριοποιείται η κοινωνία, τότε δεν υπάρχουν κοινωνικά δίκτυα, δεν είναι ελκυστική περιοχή, δεν λειτουργεί, δεν εξελίσσεται και η οικονομία. Όλοι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η οικονομική άνθηση πολλών περιοχών εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ανάπτυξη του πολιτισμού. Η επένδυση στον πολιτισμό είναι και αυτή η οικονομική ανάπτυξη και αυτό το έχουν δείξει όλες οι μελέτες. Άρα αυτή η ανάπτυξη των ψηφιακών κινηματογράφων είναι σχετικά χαμηλού του κόστους κάνει πολύ ελκυστικότερες περιοχές, η σχέση κόστος-οφέλους είναι καλή, ε, προωθείται οικονομική ανάπτυξη και σας καλώ στην εκλογική μου περιφέρεια για να το δείτε στην πράξη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αλλάζει, πρέπει να πω, την όλη δυναμική της ανάπτυξης περιοχής σχόλια από μένα και υπό την ιδιότητά μου του σκιώδου και έχω παρακολουθήσει αυτή την ε, ε, ψυχική ανάπτυξη. Αυτό που είπε για την τυποποίηση ο κ. Κρότσπα είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι βεβαίως ε, μέρος του Εβραίου, του, της ευρείας εντολής που έχουμε για το θέμα της πολιτικής των τυποποίησεων. Από την άλλη πλευρά το κόστος θα συνεχίσει να μειώνεται. Έχουμε δει το κόστος ε, ε, αντικειμένων όπως κάτι έγινε εδώ η, ε, εκρήγνεται η αντιπρόεδρός μου, ανακυκλώνει και κάνει θόρυβο. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε δει το κόστος αντικειμένων όπως η προβολής ε, να πέσουν, να πέφτει ε, εντυπωσιακά. Υπάρχει άμεση σχέση ανάμεσα στον όγκο των συναλλαγών και την διαθεσιμότητα αυτής της τεχνολογίας. Επίσης, ο κ. Κρότσμαν αναφέρει την επόμενη φάση της τεχνολογίας, γιατί ε, μιλάμε τώρα για τον τρισδιάστατο κινηματογράφο ψηφιακής τεχνολογίας 3D, γνωρίζουμε τι σημαίνει αυτό και καθώς ο κόσμος συνηθίζει πολύ υψηλή ποιότητας μεγάλες οθόνες τηλεόρασης γιατί και το κόστος ε, της, ε, των τηλεοπτικών συσκευών μειώνεται, η εμπειρία του να πηγαίνει στον κινηματογράφο με μεγάλες οθόνες πρέπει να ενισχυθεί. Όλα αυτά είναι στα πλαίσια μιας ανταγωνιστικής διαδικασίας. Επιπλέον θεωρώ ότι όλοι είμαστε ευαίσθητοι για το πόσο φθάνει ο κινηματογράφος σε διάφορες περιοχές και πράγματι ε, μπορεί μια τεχνολογία τύπου τηλεοπτικού να επιτρέπει να παρουσιάζει κανείς ε, ένα θέαμα σε μικρά κροατήρια γιατί έχουμε δει και την τεχνολογία του home cinema που ισχύει, που εφαρμόζεται παντού, να είναι χρήσιμη και εδώ. Επίσης έχουμε δει επιτυχημένα ε, πειράματα με κινητό κινηματογράφο, ασύρματο κινηματογράφο, όπου, περιοχές όπου ο καιρός είναι καλός. Είναι μια πολύ πιο ενδιαφέρουσα κοινωνικά ε, εκδήλωση αυτή. Όπως και σε πολλούς άλλους τομείς, θεωρώ ότι και εδώ η εξέπτωση η εξέλιξη της ψηφιακής τεχνολογίας θα προσφέρει πολλές πολύ περισσότερες δυνατότητες, μια πολύ διαφοροποιημένη αγορά και θα έχει ο κόσμος τη δυνατότητα να κινηθεί με ψηλή ποιότητα σε μικρότερη κλίμακα, πολύ μικρότερη από το παρελθόν. Και άρα Ας προσπέξουμε να μην ε, επιβάλλουμε μεγάλες βαρύγδουπες λύσεις σε κάτι. Να δούμε απλώς τι συμβαίνει και να ενθαρρύνουμε αυτή την ποικιλομορφία. Ωραία. Τώρα ο εκπρόσωπος της Κομισιόν είναι εδώ. Ε, κάτι θέλετε να πείτε είστε υπεύθυνο για το θέμα αυτό και κατόπιν θα δώσω πάλι το λόγο στον εισηγητή τον κύριο Κρότσμαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Κομισιόν θέλει να ευχαριστήσει τον εισηγητή και την Επιτροπή ΙΜΚΟ για μια θετική προσέγγιση του θέματος, αλλά και για τις χρήσιμες προτάσεις τους. Συμμεριζόμαστε απόλυτα τις απόψεις αυτές. Θα χρησιμοποιηθούν και στην Επιτροπή Πολιτισμού σε δύο λεπτά θέλω να σας ενημερώσω για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις. Η Κομισιόν είναι έτοιμη να ε, ξεκινήσει το δεύτερο πρόγραμμα στήριξης της ψηφιοποίησης τις επόμενες εβδομάδες. Θα, δημοσιευτεί, θα δημοσιευτούν οι προτάσεις του Συμβουλίου και το πρόγραμμα Media 2007 Έχουμε προβλέψει 2 εκατομμύρια ευρώ φέτος για αυτό το νέο πρόγραμμα. Όσον αφορά την ανησυχία των εργαζομένων στον χώρο του κινηματογράφου για μια πιθανή μείωση του προγράμματος Media στο μέλλον. Όπως γνωρίζετε, δεν θα συμβεί αυτό. Ήδη η Κομισιόν μέσω ε, ε, του Προέδρου Μπαρόζο έχει ε, εκφράσει την επιθυμία της όχι μόνο να διατηρήσει το πρόγραμμα αλλά και να το ενισχύσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε όλους όσοι πήραν το λόγο. Κύριε Κρότσμαν, θέλετε να ελέγξω το χρονοδιάγραμμα που έχουμε και μετά να κλείσουμε. Λοιπόν, έχουμε ήδη το σχέδιο της έκθεσής σας. Μιλάμε για προθεσμίες ε, Υποβολή τροπολογιών 5 Μαΐου, μελέτη των τροπολογιών και ψηφοφορία εδώ στις 25 Μαΐου, η Επιτροπή Πολιτισμού στις 15 Ιουνίου, ο κύριος Μπόρης είναι εκεί ο εισηγητής και θα πάμε στην Ολομέλεια της 4ης Ιουλίου. Λοιπόν, θέλετε να ανακεφαλαιώσετε. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους προλαλήσαντες για τις παρατηρήσεις τους, στα σχόλια. Ε, όλοι ξέρουμε ότι είμαστε πάντοτε υποποίηση χρόνου και δεν μπορούμε να συμπεριλάβουμε τα πάντα στο σχέδιο έκθεσης, οπότε βασιζόμαστε και στις τροπολογίες. Εγώ έχω το αγγλικό κείμενο και λέει rural areas. Είναι οι, περιοχέ οι περιοχές οι, οι, της υπέστρου, οι ύπεθρος δηλαδή, αγροτικές περιοχές βασικά. Το εννοώ και εγώ. Εννοώ την υπεθρό να βοηθήσουμε δηλαδή τις αγροτικές περιοχές όπου το σινεμά πρέπει να γίνει ένα γεγονός. Ε, ένα ενδιαφέρον, μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Αυτή λοιπόν η ψηφιοποίηση συνήθως χρηματοδοτείται από τις μεγάλες εταιρείες παραγωγής όμως και οι μεγάλοι παραγωγοί και οι μεγάλοι διανομή δραστηριοποιούνται στα αστικά κέντρα. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε την Ήπεθρο, γι' αυτό πρέπει να προωθήσουμε την ψηφιοποίηση και εκεί. Δεν είναι μόνο κινηματογραφικές ταινίε, αλλά και άλλα πράγματα μπορούν να μεταδοθούν ψηφιακά. Γι' αυτό είπαμε πρώτον, τα πρότυπα είναι σημαντικά, όμως δεν θέλουμε μονοπόλιο, αλλά ανοιχτή αγορά και επίσης να δώσουμε τη δυνατότητα σε ε, μη περιοχές να υποφεληθούν των εκδηλώσεων αυτών, να υποστηρίξουμε τις μη αστικές περιοχές. Βεβαίως το μέλλον ανήκει στην, ε, στις μεταδόσεις ε, HD, υψηλής ε, ευκρίνειας. Αυτό είναι αναμφίβολο. Σε ευχαριστώ λοιπόν για τις παρατηρήσεις σας και θα τις λάβω υπόψη μου στην τελική έκδοση της ε, γνωμοδότησης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κρότσμαν και εγώ. Νομίζω τώρα ε, ήδη σήμερα μάλλον μεταδιδόμαστε μέσω ίντερνετ, μέσω web stream, όχι σε τρισδιάστατη μορφή ακόμα. Λοιπόν, οι ψηφοφορίες θα αρχίσουν ακριβώς στις 10, οπότε διακόπτουμε για λίγο, μέχρι ότου πάρουν όλοι τις θέσεις τους, ολοκληρωθούν οι κατάλογοι ψηφοφοριών και στις 10 πριν να αρχίσουν οι ψηφοφορίες θα κάνω και κάποιες ανακοινώσεις. Ωραία. Σας καλωσορίζω όσους ε, ήρθατε, όσοι ήρθατε για την ψηφοφορία. Λίγη ησυχία παρακαλώ. Εάν τακτοποιείτε τον ε, κατάλογο των ψηφοφοριών, μπορείτε να το κάνετε εκτό αίθουσας, για να μην έχουμε τόση φασαρία, πριν ξεκινήσουμε και τώρα που είμαστε πολλοί, μπορώ να κάνω μερικέ σύντομε ανακοινώσει, ιδίω όσον αφορά τη συνεδρίαση των συντονιστών εχθέ. Uh, Λοιπόν, εχθέ συνεδρίαση οι συντονιστέ. Παρακαλώ ησυχία, λέει ο πρόεδρο. Παρακαλώ ησυχία στην αίθουσα. This is a very small room. Είναι μικρή αίθουσα αυτή και Παρακαλώ ε, συζητήσεις ε, έξω. Είναι χαμηλοτάβανα κιόλα και ενισχύονται οι θόρυβοι. Λοιπόν, τη Δευτέρα συνάντησα, στο, ήμουνα στο, είχα πάει στο Όσλο και συνάντησα τέσσερις υπουργούς και μάλιστα και τον Υπουργό Εμπορίου και έλαβα μέρος και στην ε, πρώτη συνεδρίαση της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για, του ΕΟΧ ΕΟΧ, Ευρωπαϊκή Ένωση, και συζητήσαμε πολλά θέματα της εσωτερικής αγοράς με τους νορβηγούς ε, ομολόγους, ε, ε, βουλευτές, υπουργούς και ενδιαφερόμενες ομάδες, ενώσεις κλπ οι Νορβηγοί πιστεύουν ότι το έργο αυτό της δικής μας Επιτροπής είναι πάρα πολύ σημαντικό και επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η Νορβηγία είναι πολύ δυναμικός εταίρος στην ε, ενιαία αγορά. Ευχαριστώ ιδίως τον κύριο Τρασκόφσκι, ο οποίος δεν είναι εδώ σήμερα γιατί συμμετέχει στις ε, τελευταίες συναντήσεις στο Spitzbergen της μικτής κοινοβουλευτικής αυτής ε, διάσκεψης και έχει πάει πολύ βόρεια κοντά στον ακτικό κύκλο για να συζητήσει μαζί με την κυρία Στάιλερ τα θέματα της εσωτερικής αγοράς εκ μέρους μας. Κάλεσα λοιπόν ε, τον Υπουργό Βιομηχανίας και Εμπορίου στις Βρυξέλλες ε, τον κύριο Γκίσκεϊ να έρθει να μας μιλήσει, να απαντήσει στα ερωτήματά σας. Μου είπε ότι θα ενδιαφέρεται ιδιαίτερα να μιλήσει ως επισκέπτη στην Επιτροπή μας. Τώρα, όσον αφορά τις αποφάσεις των συντονιστών εχθές, τα μέλη θα λάβουν βεβαίως ένα γραπτό αντίγραφο των τελικών αποφάσεων. Ορίσαμε εισηγητές ε, ορίσαμε, ε, κάναμε την κατανομή γνωμοδοτήσεων. Η Οικονομική Επιτροπή θα αναλάβει ε, το, την πρόταση καθολικής φορολογικής βάσης. Η Άλντε έχουμε μία σημαντική νέα πρόταση για, τις, για τα στεγαστικά δάνεια, υποθήκες κλπ. Αυτό θα γίνει με, στο πλαίσιο ενισχυμένη συνεργασίας με την ΕΚΟΝ σε θέματα καταναλωτών. Ε, το ΕΛΚ θα το κάνει αυτό για τις ε, επίλυση εναλλακτική, διαδικασία επίλυσης διαφορών πάλι ενισχυμένη συνεργασία με την νομική υπηρεσία. Αυτό θα πάει στην Άλντε προς μίας συνεκτική ευρωπαϊκή προσέγγιση συλλογικών προσφυγών. Αυτό θα γίνει μαζί με την νομική και Οικονομική Επιτροπή, οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες θα το κάνουν, το μέλλον του ΦΠΑ, το ΕΛΚ και αθλητισμός και Ευρώπη πάλι το ΕΛΚ. Αυτά είναι τα βασικά θέματα. Οι συντονιστές συμφώνησαν επί ενός προσωρινού προγράμματος ακρόασεων. Το, η πιο σημαντική ακρόαση είναι για τις δημόσιες προμήθειες. Η σκληρά εργαζόμενη συγγήτρια, κυρία Ρούλε, θα το αναλάβει αυτό στις 24 Μαΐου. Και ε, οι άλλες τρεις ακροάσεις είναι η αμοιβαία αναγνώριση ε, ε, των υπηρεσιών κυρία Χάνσεν, online χαρτοπέγνιο και τυχερά παιχνίδια, η τρίτη ακρόση. Επίσης, μία αντιπροσωπεία δική μας θα επισκεφθεί την Πολωνία 17-19 Μαΐου. Έχουμε πολύ καλή στήριξη της οργάνωσης αυτή από τους Πολωνούς συναδέλφους. Μπορούν και άλλες χώρες να συμμετάσχουν βεβαίως και δύο άλλα ακόμα σημεία. Πρώτον, για την επιτροπολογία συμφωνήσαμε να μην αντιταχθούμε στις ε, δύο σημαντικές ε, οδηγίες επιτροπολογίας, μία για τα μηχανοκίνητα οχήματα. Όμως, προσέξτε ότι η Κομισιόν έχει τώρα συμφωνήσει για τις προδιαγραφές ασφαλείας στα ρολά παρασύρων. Ε, αυτό άπτεται σεμάτων ασφαλείας των καταναλωτών. Λοιπόν, έχει συμφωνήσει, έχει περάσει μια συμφωνία και τώρα υπάρχουν σαφώς προδιαγραφές ασφαλείας που ισχύουν για τα ρολά, τα ρολά στα παράθυρα. Και Τέλος, οι συντονιστές συμφώνησαν ότι θα ξεκινήσουμε διαβουλεύσεις με το Συμβούλιο για να προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε μια πρώτη συμφωνία για την οδηγία δικαιωμάτων καταναλωτών. Ο πρώτος τριμερής διάλογος έγινε χτες με τον εισηγητή, τους κοιόδης εισηγητές και ε, κάναμε τα πρώτα βήματα, πιστεύω, για να βρούμε μια λύση και η Επιτροπή μας συμφώνησε να διαγράψει μια στρατηγική την οποία θα μελετήσει το Συμβούλιο και θα συνεχιστεί όλη αυτή η διαβούλευση τις επόμενες τρεις εβδομάδες. Είχαμε επίσης έναν άτυπο τριμερή διάλογο για την ετικετοποίηση κλωστοϊφαντουργικών, έξεση του κ. Μάντερς και πιστεύω ότι προχωρήσαμε και σε αυτό. Περιμένουμε όμως την τελική απόφαση. Αυτά είναι προς ενημέρωσή σας τους βασικούς φακέλους. Τυχόν ερώτηση. Όχι. Πολύ ωραία. Προχωράμε στις ψηφοφορίε. Έχουμε αρκετές νομοδοτήσεις που πρέπει να διευθετήσουμε και η πρώτη είναι η γνωμοδότησή μας για την ένβη, για τα φωσφορούχα και φωσφορούχα συστατικά στις, στα πολυπαντικά οικιακής χρήσης. Ο κύριος Ταραμπέλα έχει κάτι να μας πει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με λίγα λόγια την γραμματεία της ΣΥΜΚΟ να την ευχαριστήσω την Ζούλια Δαρνάκ για την σημαντική εργασία και το επικοδηματικό πνεύμα με τον κυρία Σαρτόρι Ρούλε, κύριο Κρόιτσμεν και Φόξ ε, συνεργάστηκα πολύ καλά μαζί τους ε, και πετύχαμε μια πολύ καλή συμφωνία. Να συνοψίσω σε τέσσερα σημεία, επιτρέψτε μου, δεν μπόρεσα να πω και πολλά πράγματα γι' αυτό. Με όλες τις ομάδες ε, συμφωνήσαμε για τις ετικέτες για τα απορριπαντικά, τα οικιακά, μετά από συμβασμό δεν ναι, θα πω λεπτομέρειες, θα μακρηγορούσα και ακόμα τρεις σημαντικές της 26, το greenwashing, το πρασινοπλήσιμο, ακριβώς ε, γιατί ε, με, υπέρ του περιβάλλοντος μέτρα είναι ακριβώς ένα σεβασμός απέναντι στην νομοθεσία που θα ισχύσει το 33 την απαγόρευση φωσφορούχων ενώσεων στα απορριπαντικά και το έχει κοινώ καταθέσει αρκετές ομάδες και έτσι ξεφύγαμε από το 0,5% ή τόσα γραμμάρια που ήταν στήρα συζήτηση και ε, από τις ζημίες προκαλούνται οι φωσφορικέ ενώσει. Ε, καταργήσαμε αυτό με τις φωσφορικέ ενώσει και η Γαλλία, α πούμε, είναι μια χώρα που αυτή η νομοθεσία από το 2007 εφαρμόστηκαν κανένα πρόβλημα με την νομοθεσία αυτή. Και επίση το επόμενο για τα υγρά απορριπαντικά, για τα πιάτα και η κυρία Ρούλ υποστήριξε επίση τα ίδια με την απαγόρευση αυτή κατά την ε, ήταν δική μου άποψη, δεν το συμμερίστηκαν όλοι, δεν υπάρχει καμία εναλλακτική λύση αποτελεσματική σήμερα, γι' αυτό περιμένουμε το 2014 και μια μελέτη από την Επιτροπή να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε, αν θα απαγορεύσουμε ή όχι στο μέλλον αυτά, αλλά προ στιγμή δεν υπάρχει κανένα υποκατάστατο που να μα ικανοποιεί τουλάχιστον στα απορριμπαντικά για τα πιάτα τα υγρά, με φωσφορικέ ενώσει ή για καθαρά πιάτα θα πρέπει να έχουμε υψηλότερη θερμοκρασία, είτε διάρκεια πλησίματο και αυτά προκαλούν όμω προβλήματα. Εντάξει, αυτά θα σα πω, δεν έχω τίποτα να προσθέσω. Σα ευχαριστώ για την προσοχή που μου αφιερώσατε. Ευχαριστώ κύριε Ταραμπέλα. Να αρχίσουμε την ψηφοφορία. Να ελέγξουμε καταρχά τι παρουσίες, αν χρησιμοποιήσουμε ηλεκτρονικέ κάρτε. θα τι χρησιμοποιήσουμε μόνο αν υπάρχει κάποια αμφιβολία. και η γραμματεία θα μου κάνει εγκαίρως ένα σήμα αν χρειάζεται. Λοιπόν, τροπολογία 1. Υπέρ, κατά, δηλαδή 23, τροπολογία 23. Δεκτή. Άρθρο 2, τροπολογία 4 του εισηγητή υπέρ, κατά, απο, ε, δεκτή. 24 του κυρίου Κρότσμαν και άλλων υπέρ, κατά, δεκτή. Τροπολογία 4α με προφορική τροπολογία του εισηγητή. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Οπότε καταπίπτει το τροπολογία 6. Τροπολογία 25 δεν ψηφίζεται. Τροπολογία 26 και πάλι με την προφορική τροπολογία του εισηγητή υπέρ κατά αποχές δεκτή. Προχωρούμε στην 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 14. Η τροπολογία 27 έχει αποσυρθεί. Πάμε στη 10 του εισηγητή υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 28 Κύριε Ρούλε, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 29 με ξεχωριστή ψηφοφορία σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος, πρώτο μέρος ψηφίζουμε. Έχει αποσυρθεί, έχει αποσυρθεί, συγγνώμη λέει ο πρόεδρος. Το δεύτερο μέρος, το δεύτερο τμήμα της 29 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 5 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τώρα προχωράμε στα παραρτήματα. 32 ε, Ρούλε. Ρούλε. Εδώ είναι ανοιχτή ψηφοφορία. Παρακαλώ ψηφίστε. Τροπολογία 32. Έληξε ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Α, 33 υπέρ. Κατά αποχές εκτή. Συμβιβαστική 1. Παράρτημα 7 υπέρ κατά, αποχές, δεκτή. Πάμε στα εκτιμώντας τώρα. Εκτιμώντας 1, τροπολογία 1, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 14, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 15, υπέρ, κατά, Απορρίπτεται 16 εκτιμώντας 2 με προφορική τροπολογία. Υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 17 της κυρίας Ρούλε, υπέρ. 17 υπέρ, κατά, άποχες, απορρίπτεται. 18 υπέρ, κατά, δεκτή. 2 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 19 ρούλε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 20 υπέρ κατά αποχές δεκτή 21 υπέρ κατά δεκτή 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή και 22 υπέρ κατά, αποχές, δεκτή. Θα κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τελική ψηφοφορία στο σχέδιο έκθεση. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. 32 υπέρ, 3 κατά, 2 αποχές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Ταραμπέλα. Um, Τώρα περνάμε στην επόμενη γνωμοδότηση που αφορά πρόταση για Deposit Guarantee Schemes. Η κυρία Ροϊκοβά Ρόιτχοβα είναι η συγγήτρια. Θέλετε να πάρετε το λόγο πριν την ψηφοφορία, κυρία Ρόιτχοβα. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τους σκιώδης. Έγιναν 82 τροπολογίες υποβλήθηκαν και μέχρι το τέλος προσπάθησα να καταλήξω γιατί θεώρησα ότι είναι σημαντικό μια γνωμοδότηση της Επιτροπής μας να έχει ευρεία στήριξη. Έχουμε μία προφορική τροπολογία και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να στηρίξουμε τους καταναλωτές μετά την οικονομική κρίση. Δεν νομίζω ότι έχουμε χρόνο να σας εξηγήσω το περιεχόμενο των συμβιβασμών, όμως θέλω να επισημάνω ότι την τελευταία ημέρα υποβλήθηκαν τροπολογίες των σοσιαλιστών που οδήγησαν σε μια αλλαγή που δεν υπάρχει τους φακέλους σας. Η κυρία Γκέπχαρτ θα τα εξηγήσει. Είναι ο συμβιβασμό υπαριθμών 14, τον οποίο στηρίζω. Είναι μια τεχνική βελτίωση, θεωρώ. Λοιπόν, να το συζητήσουμε αυτό όταν φτάσει η στιγμή να το ψηφίσουμε. Οπότε θα δώσω τότε το λόγο στην κυρία Γκέπχαρτ ακριβώς πριν ψηφιστεί αυτό. Οπότε προχωράμε. Ξεκινάμε με την τροπολογία 40 του άρθρου 2. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Η 7 αποσύρεται, 41 υπέρ κατά εγκρίνεται. Η 8 το αντιστοίχο μέρος που είναι στον κατάλογο των ψηφοφοριών υπέρ κατά εγκρίνεται. Και το δεύτερο μέρος αποσύρεται. Πάμε στο συμβιβασμό. Συμβαστική τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Περνάμε στο άρθρο 45, τροπο, προφορική τροπολογία του εισηγητή στο τέλος του, ψηφου, του καταλόγου υπέρ κατά εγκρίνεται. 10, τροπολογία 10 της εισηγήτριας υπέρ κατά εγκρίνεται. 46 της κυρίας Στάιλερ υπέρ κατά εγκρίνεται επίσης. Τώρα φτάνουμε στο στη συμβαστική τροπολογία υπάρχουν 2 και τα αντίστοιχο εκτιμώντα θα τα ψηφίσουμε μαζί. Υπέρ των δύο αυτών συμβαστικών τροπολογιών κατά σαφώς εγκρίνεται. Κατόπιν 49 της κυρία Στάιλερ. Ψηφίζουμε. Γιατί 49 ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας. Και απορρίπτεται με 26 κατά 10 υπέρ. Η 50 της κυρίας Στάιλερ υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3 υπέρ. Κατά επίσης εγκρίνεται. Περνάμε στην 59 λοιπόν υπέρ. Κατά Απορρίπτεται. Η 60 της κυρίας Στάιλερ. Υπέρ. Α, έχει αποσυρθεί φεωνάζουν. Έχει αποσυρθεί. Η 61. 61. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η κυρία Γκέπαρτ για το συμβαστική 14. Ευχαριστώ είναι προφορική τροπολογία της κυρίας Ρόιτερ που μας είχε ανακοινώσει και μάλιστα είναι το τελευταίο, τελευταίο σημείο λέει ότι α, επιστοτικά ιδρύματα τα οποία λειτουργούν υπό διαφορετική επωνυμία. Η πρώτη διατύπωση ήταν αφιλεγόμενη και μπορούσε να οδηγήσει σε παρανοήσεις. Ε, οπότε βελτιώθηκε αυτή η διατύπωση ε, και καλύπτει ε, χρηματοπιστωτικά ειδήματα τα οποία λειτουργούν με διαφορετική επωνυμία. Οπότε, έχουμε προφορική τροπολογία η οποία είναι στο τελευταία σελίδα του καταλόγου ψηφοφοριών και λέμε ότι, και το διαβάζω για να το ελέγξουμε ότι όλοι οι πιστοτικοί οργανισμοί των κρατών μελών που εφαρμόζουν αυτές τις διατάξεις δεν, δεν μπορούν να επιτρέψουν πιστοτικούς οργανισμούς να βγήσουν με διαφορετικό brand, με διαφορετική επωνυμία. Οπότε, ψηφίζουμε υπέρ της 14 κατά εγκρίνεται. Πάμε στην συμβαστική 4 υπέρ κατά εγκρίνεται. Περνάμε και η 15 έχει αποσυρθεί, οπότε πάμε στην 64 της κυρίας Στάιλερ. Ψηφίζουμε. 64 της κυρίας Στάιλερ. Ψηφίζουμε για την 64. Πέρας. Απορρίπτεται. Πάμε στην 65. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 66. Υπέρ. Κατά. Επίσης απορρίπτεται. Περνάμε στο άρθρο 9. Η 67. Υπέρ Νομίζω θα αρχίσει η ψηφοφορία για την 67 κυρίου Σβάμπ. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 22 υπέρ, 15 κατά. Η 16 δεν θα τεθεί σε ψηφοφορία. Η 68 της εισηγήτριας υπέρ. Ψηφίζουμε για την 68. Πέρας εγκρίνεται 19-17. 69 δεν ψηφίζουμε, είναι γλωσσική αλλαγή. 70. Ψηφοφορία για την 70. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 17. Το αντίστοιχο μέρος. Ψηφίζουμε για τη 17 ο πρώτο μέρος. Πέρας. Επίσης εγκρίνεται. Η 17, δεύτερο μέρος, έχει καλυφθεί από το συμβιβασμό. Πάμε στη 18 της κυρίας Ρόιτοβα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 71 Σφάμπ. Ψηφίζουμε για την 71 του κύριου Σφάμπ. Πέρας. Επίσης εγκρίνεται. Περνάμε στη 19 της εισηγήτριας, η κυρία Ρόιτοβα, δηλαδή, ψηφίζουμε για τη 19. Πέρας. Επίσης εγκρίνεται. Περνάμε στη συμβαστική υπαρχημόν υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Και μετά στην 21 της κυρίας Ρόιτοβα. 21 της κυρίας Ρόιτοβα. Ο κύριος Γκέπαρτ. Κυρία Γκέπαρτ. Θέλουμε τροπολογία σε δύο τμήματα, το, το συμφωνήσαμε με τις ομάδες. όπου δίνουμε τη δυνατότητα σε αυτή την περίπτωση ο καταθέτης να αποσύρει τις καταθέσεις του χωρίς ποινή, λαμβάνοντας τα, τους τόκους που δικαιούται κλπ. Είμαστε αντίθετοι στη συμπερίληψη του όρου sufficient, επαρκής. Ε, και είμαστε υπέρ του δεύτερου τμήματος κατά του πρώτου. Um, uh, ε, τώρα, τεχνικά δεν έχει υποβληθεί εγκαίρο το αίτημα, αλλά αν οι άλλε πολιτικέ ομάδε δεν έχουν αντίρρηση, να το να κάνουμε χωριστή ψηφοφορία. Δεν βλέπω αντιρρήσει. Προτείνω λοιπόν να ψηφίσουμε συνολικά στο για το κείμενο χωρίς τον όρο sufficient και μετά πρώτα λοιπόν χωρίς το sufficient. Ποιοι είναι υπέρ. Όλο το κείμενο. Ψηφίζουμε για όλο το κείμενο χωρίς το sufficient. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Οπότε ψηφίζουμε τώρα για τη λέξη sufficient, επαρκής. Χώρισα, χώρισα τη, ψηφοφορία. Εγκρίθηκε, εγκρίθηκε. Λοιπόν, αρχή της ψηφοφορίας για το sufficient. Ή, ε, επαρκεί ή δεν επαρκεί. Για να δούμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην συμβιβαστική 12. Υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Οπότε, η 23 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Η συμβαστική 7 υπέρ, κατά, επίσης εγκρίνεται. Η 76 της κυρίας Στάιλαρ υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Η συμβαστική 8 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Και πάμε στα Παραρτήματα. 26 της εισηγήτριας. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 27 της εισηγήτριας. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 28. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 29 υπέρ κατά εγκρίνεται. Η 77 καταπίπτει, η 30 δεν ψηφίζεται, η 78. Η κυρία Στάιλερ βέβαια στο αντίστοιχο μέρος υπέρ κατά εγκρίνεται. 78 το αντίστοιχο μέρος καταπίπτει, οπότε περνάμε στη 79-80, φτάνουμε στην 31 της κυρίας Ρόντγοβα υπέρ κατά ψήφι, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 13 υπέρ κατά εγκρίνεται. Η 33 της κυρίας Ρότοβα υπέρ κατά εγκρίνεται. Η 34 της κυρίας Ρότοβα υπέρ κατά εγκρίνεται. Η 82 καταπίπτει. Η 35 της κυρίας Στάιλερ υπέρ κατά εγκρίνεται. Η 1 της κυρίας Ρότοβα υπέρ κατά εγκρίνεται. Η συμβιβαστική 9 υπέρ, κατά, εγκρίνεται σαφώς. Η 10, συμβιβαστική 10 υπέρ, κατά, επίσης εγκρίνεται σαφώς. Φτάσαμε λοιπόν στην αιτιολογική σκέψη 32, τροπολογία 5. Ψηφίζουμε για το 5. Πέρας. Εγκρίνεται λοιπόν. Η 6. Ψηφίζουμε για την 6. Πέρας. Εγκρίνεται επίσης. Και τέλος, τροπολογία 39 του κυρίου Σμιτ υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Οπότε περνάμε τώρα στην τελική ψηφοφορία, η οποία θα γίνει ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε για την τελική γνωμοδότηση. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Οπότε εγκρίνεται 34 υπέρ, 0 κατά και 3 αποχές. Ευχαριστούμε την κυρία Ρότοβα πολύ θερμά. Θέλω να, να ευχαριστήσω θερμά το βοηθό μου. Ήταν εξαιρετικός. Um. Ωραία. Προχωράμε τώρα στη δική μου γνωμοδότηση και θα σας την παρουσιάσω. Το φαντάζομαι να έχετε αντίρρηση. Καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσω τον σκιώδη συγητή, τους σκιώδης εισηγητές, διότι δέχτηκα τις περισσότερες τροπολογίες τους, διότι πιστεύω ότι προσθέτουν αξία. Υπάρχουν πολύ λίγα τμήματα στα οποία διαφωνώ, λίγα σημεία. Ε, πιστεύω γενικά ότι θα υποστηρίξετε αυτή τη γνωμοδότηση, δεν χρειάζεται να μακρηγορήσω και ας προχωρήσουμε απευθεία στην ψηφοφορία. Ωραία. Λοιπόν, τροπολογία 1 γκρέχ, υπέρ κατά δεκτή. Συμβιβαστική ένα, υπέρ κατά αποχές δεκτή. Γι' αυτό προχωράμε στο 4. Κόρχολα, κοράτσα μπίλτ υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 5. Βάσκερμπερ ε, υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 10. Τροπολογία 10 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή και 11 υπέρ κατά δεκτή, οπότε θα γίνει νέα παράγραφος. Συμβαστική 3 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 13. Βάσκερμπερ, υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 14 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 15 Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 16. Γκρέχ. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 17. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 18. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 19. Υπέρ, κατά, αποχές δεκτή και ε, σύμφωνο ε, να μετακινηθεί ε, πριν από την παράγραφο 3. 20 επίσης δεκτό, ε, απολυγία 21 δεκτή, ε, απολυγία 22 με προφορική τροπολογία που βλέπετε στον κατάλογο εδώ υπέρ, κατά, αποχές δεκτή, 22 καταπίπτει, 23 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 24 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 25 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 26 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ψηφίζουμε την, τροπολο... την ε, γνωμοδότηση ηλεκτρονικά στο σύνολο άρχεται ψηφοφορία. Έληξε η ψηφοφορία. Ευχαριστώ για την ε, πιστική σας υποστήριξη. Πρέπει λοιπόν τώρα να την υποστηρίξουμε έναντι της Επιτροπής Βιομηχανίας. Και έχω και τη δεύτερη γνωμοδότησή μου τώρα για τη στρατηγική ε, Ευρώπη 2020. Ήταν πιο περίπλοκο εδώ το ζήτημα και ορισμένε τροπολογίε δεν μπόρεσα να τι δεχτώ, διότι θα, και θα πρέπει να τι ψηφίσουμε. Γενικά πιστεύω ότι έχουμε συμφωνήσει ε, στους, ε, συμβιβαστικέ. Ξέρω ότι οι πράσινοι θέλουν να παρουσιάσουν προφορικές τροπολογίες. Αυτό εξαρτάται από το αν τα άλλα, ε, ε, οι άλλες ομάδες το δεχτούν. Ο κύριο Φαμπ. Βλέπω ότι η τροπολογία του Όλε Σμιτ του προβλέπει στο 1α να μπει υποστηρίζει και ενθαρρύνει την απομάκρυση των υφισταμένων προσκομμάτων στην εσωτερική αγορά. Μου εξηγείτε γιατί είσαστε εναντίον αυτής της προσθήκης. Δεν είμαι καθόλου εναντίον, λέει ο πρόεδρος αλλά σας θυμίζω ότι υπήρχε ένα σημείο τη Κομισιόν για το εξωτερικό εμπόριο μέσα στα πλαίσια της στρατηγικής 2020. Εγώ πιστεύω ότι οι γνωμοδοτήσεις πρέπει να είναι πολύ σοβαρό ζήτημα, δηλαδή πρέπει να σχετίζεται το περιεχόμενο με το θέμα επί του οποίου γνωμοδοτούμε. Και πιστεύω ότι αυτό λέει κάτι προφανές ε, και δεν χρειάζεται να περιληφθεί στη στρατηγική 2020 το οποίο, ε, στρατηγική το λέει ήδη. Λοιπόν, ε, δεν έχω τίποτα εναντίον, αλλά πιστεύω ότι επικαλύπτεται από τη στρατηγική αυτή και δεν χρειάζεται. Επίσης, στην τροπολογία 9 αναφέρεται στην ανοιχτή αγορά αεροπορικών μεταφορών, που δεν νομίζω ότι εμπίπτει στη στρατηγική 2020. Ο ως πρόεδρος θέλω οι γνωμοδοτήσεις να είναι υψηλής ποιότητος και απολύτως ε, σχετικές με το αντικείμενό τους. Γι' αυτό και ήμουν πολύ αυστηρός ε, στην εξέταση των τροπολογιών. Εάν όμως ο κύριος Σμιτ ε, θέλει να ψηφιστεί η τροπολογία του, τότε θα την θέσω προς ψήφιση. Ο κύριος Σμιτ. Ε, πολύ πιστικά επιχειρήματα. Δεν θέλω δημιουργήσω πρόβλημα. Οπότε, ακολουθώ τη συμβουλή σας. Ελπίζω να είστε καλός μαζί μου κι εσείς, αφού σας κάνω αυτή την υποχώρηση. Είμαι πάντα πολύ καλός, ε, λέει ο πρόεδρος, και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που συμμετέχετε στην Επιτροπή. Η κυρία Ντεγκρίτ και εγώ κάναμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για το, την 22 άμεσες επενδύσεις που δεν νομίζω να έχει πολύ σχέση με την Ευρώπη 2020 ε, δεν μπόρεσα να την υποστηρίξω αυτή την τροπολογία, αν όμως άλλοι τη θέλουν οπωσδήποτε, ας την ψηφίσουμε εγώ χωρισμένες επιφυλάξεις. Επίσης ζήτησα ξεχωριστή ψηφοφορία για την τροπολογία της κυρίας ε, Στάιλερ εκ μέρους της δικιάς μου μας ομάδας. Γιατί υπάρχουν ακόμα ε, μερικές αμφιβολίες για τα χρηματοδοτικά αυτά μέσα, εάν θα είναι παραδοσιακά ή καινοτομικά. Από φαίνεται τα, οι καινοτομικέ χρηματοδοτήσεις βρίσκουν χρήματα έτσι, ουρανοκατέβατα από κάπου ε, από την ατμόσφαιρα, από τον αέρα. Λοιπόν, έχω ορισμένε αμφιβολίες για την πιστικότητα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. να απαντήσω, αν μου επιτρέπετε, αυτά που είπατε μόλις ε, για την 22 τροπολογία που εγώ έχω υποβάλει. Η τροπολογία αυτή 22 δεν προσπαθούσε να κρύψει μια κάποια τάση προστατευτισμού, οποιαδήποτε τάση και δεν ήθελα να αλλάξει το πνεύμα από το οποίο προωθεί τις εμπορικές σχέσεις Ευρωπαϊκή Ένωση με τον υπόλοιπο κόσμο. Απλά και μόνο σε ένα πνεύμα ανοίγματο μπορούμε να πούμε και υπεύθυνο και ρεαλιστικό πνεύμα που αποκλείει οποιαδήποτε αφέλεια και να έχουμε τη δυνατότητα για ένα εργαλείο για να γνωρίζουμε καλύτερα, να μελετάμε καλύτερα τις επιπτώσεις της άμεσες ορισμένων επενδύσεων, ξένων επενδύσεων που περιέχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διάφορους στρατηγικούς τομείς της οικονομίας μας. Το εργαλείο αυτό προτείνεται και από ορισμένου εξέχοντε επιτρόπου Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να έχουμε καλύτερη γνώση και να κάνουμε και σωστότερη και αμεσότερη διάγνωση. Ευχαριστώ. Υποθέτω, λέει ο πρόεδρο, ότι η Επιτροπή θα συμφωνήσει μαζί σα. Θα δούμε. Λοιπόν, προχωρούμε στην ψηφοφορία. Συμβιβαστική 1 υπέρ. Κατά. Να, να ελέγξουμε παρακαλώ. Η, η το, συμβιβαστική 1. 1. Συμβιβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. Οπότε προχωρούμε ε, στην, ε, στο, στην τροπολογία degree 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 5 Legrip υπέρ κατά Α, να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Παράγραφο, ε, τροπολογία 5 Legrip. Άρχεται η ψηφοφορία. Έλξε η ψηφοφορία. Δεκτή. Ο κύριο Σμιτ ευγενώ απέσυρε την τροπολογία 6 και προχωρούμε στη συμβαστική 2. Υπέρ, κατά, δεκτή. Τροπολογία 9. Σμιτ. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 3. Υπάρχει μια πρόταση των πρασίνων. Μπορείτε να μας την παρουσιάσετε και η Επιτροπή θα αποφασίσει αν τη δεχτεί ή όχι. Η κυρία Ρούλε. Ζητάμε ξεχωριστή ψηφοφορία για τη, διατύπωση εφαρμογή των ε, πνευματικών ε, δικαιωμάτων και αυτές enforcement of intellectual property rights εφαρμογή για τα, των δικαιωμάτων ε, πνευματικής ιδιοκτησίας. Μάλιστα, λοιπόν, θα ψηφίσουμε την συμβιβαστική τρία χωρίς τις λέξεις Enforcement of Intellectual Property Rights. Συμβαστική τρία, χωρίς αυτές τις λέξεις. Όλη τη συμβαστική τρία ψηφίζουμε. Ολόκληρη. Υπέρ. Α, δεν, δεν υπάρχει κάποια σύγχυση. Πρώτα θα ψηφίσουμε με την απάλληψη αυτής της ε, διατύπωσης, αυτού του της ε, τμήματος και μετά με το, τη διατύπωση αυτή για τα πνευματικά δικαιώματα. Ο κύριος Σβάμπ, από ό,τι καταλαβαίνει ψηφίζουμε τώρα με την απάλληψη αυτής της διατύπωσης. Πρώτα, ναι, ωραία. Λοιπόν, συνεβαστική τρία με τη διαγραφή αυτών των λέξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Περί πνευματικά δικαιώματα. Δεκτή. Τώρα ψηφίζουμε τη συνεβαστική τρία με τη διατύπωση ε, ε, επιβολή, ε, εφαρμογή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Με αυτή τη διατύπωση. Υπέρ. Κατά. Πρέπει. Λοιπόν, ε, θα περιληφθεί αυτή η διατύπωση. Θα περιληφθεί. Δεν θα διαγραφεί. Προχωράμε στην τροπολογία 17. Λεγκρίπ υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 14 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 15 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 24 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 26 24, 24 ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ 24, άρχεται η ψηφοφορία πέρα της ψηφοφορίας δεκτή για μία ψήφο. Πολύ ωραία κύριε Σμιτ. 26 Στάιλερ υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Ε, η συμβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 22 Λεγκρίπ υπέρ. Ηλεκτρονικός έλεγχος, άρχεται η ψηφοφορία. Το ΕΛΚ έχει μία ψήφο παραπάνω. Α, εντάξει, διορθώθηκε. Λοιπόν, πέρα της ψηφοφορίας, πάλι υπερψηφίστηκε με μία ψήφο παραπάνω. 23 Στάιλερ με προφορική τροπολογία. Σε δύο τμήματα. Έχουμε καταρχάς τη δημιουργία των ε, ομολόγων, ευρωπαϊκών ομολόγων έργου και θα, ψηφ... ψηφίσουμε. Καταρχάς για τη συμβαστική αυτή, χωρίς αυτή τη διατύπωση, η οποία λέει through the creation μέσω της δημιουργίας ευρωπαϊκών ομολόγων έργου, υπέρ, παρακαλώ, κατά, αποχές, δεκτή, και εν συνεχεία με τη, με τη συμπερίληψη των ομολόγων έργου. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Ένα λεπτό. And, uh, we now have a vote. Και τώρα έχουμε την τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote is... Έληξε η ψηφοφορία. Δεκτή. 33 υπέρ... Α, και τρεις αποχές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξή σας και τους δυο ηγητές. Πολύ ωραία. Προχωράμε στα προγράμματα εγγύσεων και δίνω το λόγο στον Αντιπρόεδρο Λουί Γκρέχ. Oh. Καταρχήν, κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις εισηγητές για την εξαιρετική συνεργασία. Όλοι μας, Πρόεδρε, είχαμε την καλή θέληση και, την, το μυαλό να προσπαθήσουμε να βρούμε κάποια ισορροπία, προσφέροντας υψηλό επίπεδο προστασίας στους καταναλωτές, αυτούς που έχουν ασφαλιστικά συμβόλαια, ενώ ταυτόχρονα δεν θέλαμε να επιβαρύνουμε ιδιαίτερα τις ασφαλιστικές εταιρείες. Βασικά, καταλήξαμε σε έναν καλό συμβιβασμό, θεωρώ, και αυτά είχα να πω με δύο λόγια. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε περνάμε στην ψηφοφορία. Για την γνωμοδότηση του κυρίου Γκρέχ. Παράγραφος 1, τροπολογία 4, Fox. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 3, Schwab και άλλοι. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 5 του Σαλβίνη καταπίπτει. Η 6 του εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Οπότε καταπίπτει του κυρίου Σμιτ, αν δεν κάνω λάθος. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Σαφώς εγκρίνεται. 22 του κυρίου Σφάπ και λοιπά υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 23 του εισηγητή ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Με 20 υπέρ 17 κατά. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 29 του εισηγητή Ψηφίζουμε για την 29. Πέρας. Εγκρίνεται με 20 υπέρ 16 κατά, συμβιβαστική 5 υπέρ κατά εγκρίνεται. Η 34 του κυρίου Σμιτ υπέρ κατά απορρίπτεται. Η 35 του κυρίου Κανθάν. ψηφίζουμε για την 35 Πέρας. Εγκρίνεται 21-14. 36 του κυρίου Σμιτ. Υπέρ. Α, ψηφίζουμε, ψηφίζουμε γιατί 36. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1 του εισηγητή υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 2 του εισηγητή υπέρ. Α, ψηφίζουμε, ψηφίζουμε για την τροπολογία 2. Πέρας. Εγκρίνεται. Σύνολο του σχεδίου γνωμοδότηση ηλεκτρονικά υπέρ. Ε, μάλλον ε, ψηφίζουμε. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται με 34 υπέρ, 0 κατά 3 αποχές. Συγχαρητήρια στον κύριο Γκρέχη. Ε, και τώρα περνάμε σε μια σημαντική ε, γνωμοδότηση του κυρίου Σαλβίνη, τον οποίο χαιρετίζω θερμά. Είναι η πρώτη σας γνωμοδότηση. Με τα χαρά θα σας δώσω τον λόγο για να μας ε, παρουσιάσετε τους συμβιβασμούς και τις τροπολογίες. Κύριε Σαλβίνη. Grazie, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ναι. Πρώτη μου φορά ευχαριστώ όλους τους ε, ε, συγγητή τη γραμματεία, τη γραμματέα και έτσι φτάσαμε σε συμβαστικές λύσεις. Σχεδόν όλοι συμφωνούν με αυτές τις συμβαστικές λύσεις εκτός από δύο-τρεις φρασούλες ε, για τους σοσιαλιστές και τους πράσινους έχουν ζητήσει σε ξεχωριστά μέρη ψηφοφορία, το δεχτήκαμε και σε άλλα διαφορετικά θέματα υπήρχαν πολύ πολύ λίγες και ελαφρές διαφορές. Βάσκα η πράσινη για να μπούμε σε λεπτομέρειες στο θέμα του δικαίωματο να ξεχνιέται κανείς, εντάξει, αλλά ήταν αρμοδιότητα της Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών, δεν θελήσαμε να μπούμε σε λεπτομέρειες στο δικό του χωράφι και νομίζω ότι όλοι μας πετύχαμε μια καλή συμφωνία και ο Μαΐου θα εξετάσει το θέμα στην ε, Επιτροπή Ελευθεριών και στο τέλο Ιουνίου ψηφορία στι Βρυξέλλε. Νομίζω ότι πετύχαμε στην καλύτερη δυνατή συμβαστική λύση, λύσεις. Ευχαριστώ για την εργασία σας. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα εξαιρετικά ενδιαφέρον και πρέπει να παρακολουθήσουμε το θέμα με τον Πρόεδρο Μπαρόζο. Έχουμε 74 ε, τροπολογίες, είναι το μεγαλύτερο πακέτο της ημέρας. Ας ψηφίσουμε λοιπόν. Συμβιβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Περνάμε κατευθείαν στην 19 του κυρίου Γκρέκ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 17 της κυρίας Γκέπχαρτ. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 16 Κρότσμαν. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά. Επίσης εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2. Υπάρχει αίτημα χωριστή ψηφοφορία από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Είναι ξεκάθαρο σε όλου σα. δεν θα σας το διαβάσω, θα δείτε γιατί θα ψηφίσουμε. Λοιπόν, πρώτο μέρος της συμβαστικής τροπολογία υπέρ, κατά, Σαφώ εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος της συμβαστική. ηλεκτρονικά, ψηφίζουμε για το δεύτερο μέρος τη δεύτερης συμβιβαστικής. Πέρας. Εγκρίνεται και το δεύτερο μέρος με 27 υπέρ. Περνάμε κατευθείαν στην τροπολογία 25, η οποία έχει συμφωνηθεί να είναι προσθήκη στον συμβιβαστική 2. Ψηφίζουμε για την 25. Πέρας. Απορρίπτεται με 21-15 του κυρίου Γκρέχ, 29 υπέρ, κατά εγκρίνεται. 30 της κυρίου Σαλντεμόζα υπέρ, κατά εγκρίνεται. 28 του κυρίου Κρότσμαν υπέρ, κατά εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στη 32 με προφορική τροπολογία που αναφέρεται στον κατάλογο ψηφοφοριών με την προφορική υπέρ κατά εγκρίνεται. Χωρίς λοιπόν την απορρίπτεται μετά. 33 ή 33. Ηλεκτρονικά. Πέρας. Απορρίπτεται. Η συμβαστική 3 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Περνάμε λοιπόν στην 42 του κυρίου Ζουβάν υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 40 Κρότσμαν, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 43 Ζουβά, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Η 51 της κυρίας Γκέπχαρτ, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 53 με προφορική που αναφέρεται εδώ στον κατάλογο, υπέρ, κατά, σαφώς εγκρίνεται. 55 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 57 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 56 με προσθήκη και ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 56. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 58 της κυρίας Αρντιμόζο υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 60 του κυρίου Βαντεκάμπ. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Η συμβαστική 7 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Και περνάμε στην 59 ως προσθήκη υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 62 υπέρ. Κατά αποχές επίσης εγκρίνεται. Η 63 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 64 ηλεκτρονικά. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 66 του εισηγητή. Ηλεκτρονικά. Πέρας. Εγκρίνεται με 20 υπέρ 17 κατά. Η 68 του κ. Ζουβάν υπέρ κατά εγκρίνεται. Η συμβιβαστική 6 σε δύο μέρη. Χωριστή ψηφοφορία ζητούν οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες. Αναφέρεται στον κατάλογο. Λοιπόν, ψηφίζουμε το πρώτο μέρος υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Και δεύτερο μέρος ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε για το δεύτερο μέρος μέρο 6, πέρας, εγκρίνεται. Περνάμε στην 71 του κυρίου Κρότσμαν. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 72 Ζουβά υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 69 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 73 ηλεκτρονικά. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 74 ζουβά υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ένα της κυρίας Γκέπχαρτ. Έχουμε φτάσει στη θεολογία σκέψη. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 5 ως προσθήκη του συμβιβαστικής 8 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 8 ως προσθήκη υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 7 του κυρίου Γκρέχ υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Η 6 της κυρίας Γκέπχαρτ υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Η 9 της κυρίας Γκέπχαρτ ηλεκτρονικά. Πέρας, εγκρίνεται. Οπότε, γίνεται ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σύνολο της γνωμοδότησης. Υπάρχει κάποιο που δεν θέλει να ψηφίσει. Πέρας ψηφοφορίας. Χάνουμε έναν, κάποιος δεν ψήφισε. Εν πάση περιπτώσει, 36 υπέρ, 0 κατά. Κύριε Σαλβίνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Οπότε σας αφήνουμε να το υπερασπιστείτε στην ε, Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Δύσκολη δουλειά. Περνάμε στην τελική ψηφοφορία που είναι μία και μοναδική και αφορά το πρωτόκολλο της Ανδόρας. Ο εισηγητή μα είναι ο κύριος Μάντερς. Θέλετε να πείτε... Όχι, απλώ να ευχαριστήσω όλους, τη γραμματεία, του Σκιώδης. Είμαστε, έχουμε προετοιμάσει πολλές τροπολογίες, αλλά τελικά το μόνο που αποφασίσαμε ήταν να πούμε ναι ή όχι και είπαμε ναι και τελείωσε. Σας εύχομαι να έχετε πάντα τόσο εύκολες εκθέσεις, κύριε Μάντερς. Μία ψηφοφορία υπέρ, κατά, Σαφώς εγκρίνεται. Οπότε, ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι, είμαστε ακριβώς στην ώρα μας. Θα σας αφήσω ε, λίγο χρόνο για να φύγουν όσοι δεν θα μείνουν στην επόμενη συζήτηση. Θέλω απλώς να σας υπενθυμίσω όσοι από εσά που δεν θα μείνετε για το υπόλοιπο του πρωινού, ελπίζω να μείνετε, αλλά αν φύγετε, ο κύριος Μπαρνιέ, ο Επίτροπος, θα έρθει κατά βάση πιθανότητα στι 3 το απόγευμα. Είναι πολύ σημαντική η συνάντησή μας μαζί του, γιατί παρουσιάζεται η πράξη ενιαίας αγοράς που θα ανακοινωθεί στις 11 από την Κομισιόν. Τώρα, είναι η πρώτη ευκαιρία που έχει το Κοινοβούλιο. Εσείς να τον ακούσετε να μιλάει για την πράξη ενιαίας αγοράς και να τον ρωτήσετε επ' αυτού. Λοιπόν, παρακαλώ να έρθετε όλοι στις 3 η ώρα στη συνάντηση με τον Επίτροπο Μπαρνιέ. Οπότε διακόπτουμε για λίγο, πολύ λίγο, όποιος θέλει να φύγει. Ας φύγει και κατόπιν θα δώσω το λόγο στην κυρία Γκέπχαρτ.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 Uh, right. We are now going to, um... πλέον, περνάμε στο επόμενο θέμα της ημερησίας διάταξης, που είναι... Give a minute For our rapporteur. So, uh... Περιμένω την, τον, την, τον εισηγητή. Κορνέλης. Good. Λοιπόν, κάνουμε την πρώτη ανταλλαγή απόψε για μια σημαντική γνωμοδότηση για τις τεχνικές προδιαγραφές που χρειάζονται για τις μεταφορές πιστώσεων και άμεσων χρεώσεων σε ευρώ και την, ε, τον, τον κανονισμό που θα τροποποιηθεί. Ο κύριος Σουάπ άλλος. Ε, το ΕΛΚ είναι... Α, λείπει ο εκπρόσωπος ε, του ΕΛΚ για τον εισηγητή. Ο κύριος Σμιτ όμως θα μπορέσει να τα αναλάβει. Ο κύριος Κάμφαντ από τους Πράσινους δεν είναι, κύριε Ριούλε θα καλύψει. Ευρωπαίοι συντηρητικοί, κανείς εδώ εθελοντής. Uh, Um, and uh, κυρία Γκέπαρτ, έχουμε μισή ώρα για αυτή τη συζήτηση και πρέπει να είμαστε σχετικά σύντομοι. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομη. Είναι και η πρώτη ανταλλαγή που κάνουμε και θα επακολουθήσουν συζητήσεις οπότε θα σας κάνω εδώ την πρώτη παρουσίαση. Η γνωμοδότηση αυτή είναι με τεχνικής φύσεως, αλλά έχει και πολιτικές επιπτώσεις, διότι θέλουμε να απλουστεύσουμε τις μεταφορές χρημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ιδίως τις διασυνοριακές μεταφορές χρημάτων και ε, όλοι οι τρόποι πληρωμής από εθνικής απόψεως μέσω λογαριασμών ε, αντικαθίσταται τώρα με το IBAN και το BIC για να μπορούν να γίνονται πιο εύκολα οι διασυνοριακές, ε, οι διακρατικές ε, μεταφορές πιστώσεων. Είναι μια, ένας ευρύτατος τομέας και σκέφτηκα πώς θα μπορέσω να αντιμετωπίσω αυτό το ζήτημα. Ε, πολλοί πολίτες μας έχουν συνηθίσει το παλιό σύστημα και κάθε φορά που γίνεται υποχρεωτική μία αλλαγή, τα πράγματα δυσκολε... τους δυσκολεύουν η προθεσμία και που έβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε πολύ σύντομες, σύντομες προθεσμίες για την επιβολή αυτών των αλλαγών. Αποφάσισα λοιπόν να προτείνω στην Επιτροπή να ακολουθήσουμε την οδό που προτείνει η Κομισιόν. Δηλαδή μετά από μια μεταβατική φάση να φροντίσουμε να ισχύουν ενιαίοι τρόποι πληρωμών μέσω IBAN και BIC. Βέβαια, θα πρέπει να, ξε... αποσαφηνίσουμε ότι οι προθεσμίες που έθεσε η Κομισιόν ε, δεν είναι καθόλου επαρκής. Δηλαδή ένας ε, μεταβατικός χρόνος ή το πολύ δύο, δύο χρόνια εδώ οι καταναλωτές πρέπει να προσαρμοστούν στις αλλαγές, να κατανοήσουν τις αλλαγές. Και βεβαίως ο πολλαψή, πολλαψήφιος αυτός αριθμός του IBAN ε, μπερδεύει ακόμα ε, τους καταναλωτές γιατί έχει 25-27 ψηφία ε, και δεν είναι τόσο δύσκολος αυτός ο αριθμός αλλά λένε βεβαίως οι περισσότεροι ε, ε, πελά, καταναλωτές ότι δεν μπορούν να το θυμούνται απ' έξω επειδή έχει τουλάχιστον 25 στοιχεία. Επίσης για τις ε, μικρές επιχειρήσεις οι οποίες ε, έχουν αυτή τη στιγμή ένα σύστημα το οποίο εφαρμόζουν και συνεργάζονται και με μικρότερες τράπεζες και αυτές οι μικρότερες επιχειρήσεις μας έχουν πει ότι θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες διότι πρέπει να αλλάξουν τα λογισμικά του συστήματα ε, και τις διαδικασίες τους. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν δυσκολίες και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Λέω λοιπόν να πούμε εντάξει, δεχόμεσα το δρόμο που προτείνει η Κομπισιόν, μία εναρμόνιση των ευρωπαϊκών τρόπων, μεθόδων μεταφοράς πιστώσεων, αλλά θέλουμε περισσότερο περιθώριο προσαρμογής. Και γι' αυτό προτείνω για την Τέλεση της μεταφοράς αντί 24 μήνες να προβλέψουμε 48 και δεν βρίσκω τις τροπολογίες μου τώρα. <laughs> Τα έχω μπερδέψει, λέει η κυρία Γκέπαρτ. Εν πάση περιπτώσει, να ζητήσουμε μία ουσιαστική παράταση των προθεσμιών για την εφαρμογή αυτών των αλλαγών για να μπορούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι να τις συνηθίσουν, να τις κατανοήσουν και να προσαρμοστούν και για να μην επιβαρύνουμε ε, τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις να εφαρμόσουν αλλαγές σύντομα και ε, χωρίς να τις έχουν ακριβώς καταλάβει. Είναι ουσιαστικές αυτές οι αλλαγές. Επίσης η τοπική αυτοδιοίκηση επηρεάζεται. Αναμφίβολα Χρειαζόμαστε λοιπόν για αυτή τη μετατροπή του συστήματος περισσότερο χρονικό διάστημα. Αυτό ε, είναι βέβαιο. Επόμενο ζήτημα είναι πώς θα ρυθμίσουμε το θέμα αυτό και δεδομένου ότι επεξεργάστηκα όλα αυτά τα ζητήματα στα αγγλικά, ε, με τη γραμματεία δεν μου έρχονται οι λέξεις στα γερμανικά, πώς θα γίνουν αυτά τα air transactions. Εδώ πρέπει να ξέρουμε ποιος πληρώνει, ποιος είναι υπεύθυνο για να... το κόστος, τη δαπάνη η οποία δημιουργείται. Εάν η Κομισιόν θέλει να επιβαρυνθούν οι καταναλωτές με αυτές τις δαπάνες, εδώ πρέπει να βρούμε μια πιο καλή ισορροπία σε αυτά τα air transactions. Επίσης, στα, στο άρθρο 18 θα προτείνω στους τομείς ε, οι οποίοι καλύπτουν ε, παράπλευρα ή δευτερεύοντα προϊόντα να δοθεί αρκετή προθεσμία ε, προσαρμογής ε, εύλογη. Διότι μέχρι το 2012, όταν μιλάμε για παράπλευρα ή συνεπαγόμενα προϊόντα, μου φαίνεται η προθεσμία είναι πάρα πολύ στενή. Και τρίτο ζήτημα είναι οι διατάξεις του παραρτήματος 1. Ένα μεγάλο μέρος των διατάξεων του παραρτήματος 1 και που εμπίπτουν στην επιτροπολογία θα προτιμούσαν να ενταχθούν στο διατακτικό με τη μορφή άρθρων, διότι είναι ζητήματα τα οποία δεν θέλω να τα αφήσω στα χέρια της Κομισιόν. Κοιτάω την Κομισιόν βεβαίως εδώ, στα μάτια. Προτιμώ να έχουμε και εμείς λέγειν επί αυτών των ε, διατάξεων. Αυτές οι διατάξεις λοιπόν στο παράρτημα 1 θα ήθελα να μπουν σε άρθρα είναι ζητήματα προσαρμογής, ζητήματα προτύπων, διαφοράς, διαφορετικών προτύπων που υπάρχουν. Εδώ πρέπει να προχωρήσουμε πολύ προσεκτικά, γιατί έχει και πάλι μεγάλη σημασία στη... για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτά λοιπόν, έτσι ως πρώτη παρουσίαση. Ωραία, σήξατε πολλά ενδιαφέροντα θέματα και πρέπει να ε, τα προσέξουμε. Ο κύριος Σμιτ, ο οποίος είναι εμπειρογνώμος σε αυτό το τομέα. Ευχαριστώ. Όπως είπε η συγγήτρια, αυτή είναι μια εξαιρετικά σημαντική γνωμοδότηση. Το ερώτημα είναι γιατί καθυστερήσαμε τόσο πολύ να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Ποιοι είναι οι λόγοι. Είναι επειδή καθυστερούμε στην αντιμετώπιση νομοθετικών ε, ζητημάτων ή επειδή οι τράπεζες καθυστερούν ε, την αλλαγή του συστήματος. 4-5 χρόνια είναι που συζητιούνται αυτές οι αλλαγές. Και όπως είπε το Κοινοβούλιο και η συγγήτρια. Ε, χρειαζόμαστε να προχωρήσουμε γρήγορα εάν θέλουμε να ολοκληρώσουμε την ενιαία αγορά. Αυτό το θέμα της ε, μεταφοράς πιστώσεων και άμεσων χρεώσεων κλπ. είναι ένα θέμα κλειδί. Δεν είμαι έτοιμο σήμερα να πω εάν ε, αυτά τα οποία προτείνει η Κομισιόν όσον αφορά τις προθεσμίες, δηλαδή είναι αποδεκτά ή όχι. Θα το μελετήσω δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν και επίσης θα ήθελα να κοιτάξω ε, τι προτείνουν οι άλλες ομάδες σε αυτό τον τομέα. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μία κοινή θέση από απόψε της Επιτροπής. Επίσης, έχω μία επιπρόσθετη παρατήρηση Ε, θα μπορούσα ίσως να μιλήσω εκ μέρους μιας αυξανόμενης μειοψηφίας. Λέγοντας ότι η πρόταση αυτή ευνοεί το χρονοδιάγραμμα των ευρωπαϊκών κρατών. Δεν ξέρω αν ο πρόεδρο συμμερίζεται την άποψή μου. Αλλά αυτό το οποίο γίνεται σήμερα στην Ευρώπη είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, διότι διαιρούμε την Ευρώπη σε μια Ευρώπη όχι μόνο δύο, αλλά ενδεχομένω τριών ταχυτήτων. Και μακροπρόθεσμα θα έλεγα ότι αυτό θα δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα στην, ευρωπαϊκή, στην ενιαία αγορά ακόμα και αν εφαρμοστεί το Europe Plus, το Europe Sin όπως είπε ο Επίτροπος Μπαρνιέ. και κατά τη δική μου άποψη και θα ήθελα να ακούσω και την άποψη συναδέλφων που δεν έχουν το ευρώ. Εγώ θα ήθελα η χώρα μου να υιοθετήσει το ευρώ, αλλά ακόμα και αν δεν είναι στην ευρωζώνη, θα πρέπει να είμαστε σε αυτό το σύστημα. Διότι ειδικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι εξαγωγές που γίνονται από τη χώρα μου γίνονται μέσω της Ευρωζώνης και η μεγαλύτερη, ο μεγαλύτερος όγκος εξαγωγών γίνεται στη Γερμανία. Οπότε βεβαίω έχουμε ένα λόγο παραπάνω να υιοθετήσουμε αυτό το σύστημα και να αποφεληθούμε από την ενιαία αγορά. Γι' αυτό λοιπόν ρωτώ την Κομισιόν, γιατί μας το κάνετε αυτό, γιατί οι εκτός Ευρωζώνης δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτές τις ε, αλλαγές, σε αυτές τις τεχνικές αλλαγές. Θα ακούσω την απάντηση και θα επανέλθω. Ο πρόεδρος ε, προέρχεται από χώρα εκτός Ευρωζώνης, ε, οπότε μπορεί να έχουμε διαφορετικές απόψεις, αλλά ας ακούσουμε και την κυρία Ρίλε. πρέπει να πω ότι δεν συζήτησα με τον σκιώδη συγητή μας μέχρι τώρα. Γι' αυτό θα είμαι πολύ, πολύ προσεκτική. Δίνω, δικαιολογώ τον κύριο Σμιτ τις επικρίσεις του και η Γερμανία χρειάστηκε πολύ διάστημα να αποσαρμοστεί και ακόμα έχει πολλά να κάνει. Εμένα πάντοτε μου λένε ότι ξέρετε δεν μπορούμε να το κάνουμε, κάνουμε τη, τη μεταφορά ή την α ή β συναλλαγή, διότι υπάρχουν τεχνικά προβλήματα. Και δεν υπήρχε προθυμία και επίσης δεν ασκήσαμε αρκετή πίεση να υιοθετηθούν αυτές οι αλλαγές. Είμαστε σε δύσκολη θέση. Πρέπει να το μελετήσω με, τους, ε, με το σκιώδη συγγητή μας, διότι δεν έχουμε ακόμα θέση, διαμορφώσει τη θέση μας ως ομάδα. Και επίσης σε εθνικό επίπεδο πρέπει να το συζητήσω, αλλά το παράπανό σας το κατανοώ απόλυτα. Το 7 τι είναι, δεν έχει. Κύριε Πρόεδρε, σύντομα σύντομα ένα σχόλιο από δικής μου πλευράς. Προέρχομαι από μια χώρα που δεν ε, χρησιμοποιεί το ευρώ. Και ορισμένοι μας αποκαλούν ευρωσκεπτικιστές, αλλά μάλλον πως είμαστε ευρωρεαλιστές και όχι ευρωσκεπτικιστές. Για μας η ιδιαίτερη σημασία για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι ακριβώς η ιδέα περί έννοιας αγοράς. Και αν ανατρέξουμε στη ξεκίνημα ε, είναι σημαντικό το ότι παρατηρούμε με διαφορετικά νομίσματα χώρες. Εντάξει, δεν θα επιμείνω σε αυτό το σημείο αλλά το σημαντικό ποιο είναι, ότι η νέα αγορά χρειάζεται κάτι περισσότερο από ένα κοινό σύστημα πληρωμών. Παρακαλώ επίσης προσέξτε εσείς την Επιτροπή για ένα σύστημα για περισσότερη γραφειοκρατία έτσι χαρτιά εδώ και εκεί και εμπόδια για τους πολίτες, ε, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ακόμα για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Εδώ θα μπορούσαμε ίσως να το συζητήσουμε με τον κύριο Μπαρνιέ σήμερα το απόγευμα θα μπορούσε να αποδειχθεί ενδιαφέρον και στη δημοκρατία της Τσεχίας. Τη βδομάδα που μας πέρασε συζητήσαμε για το Ευρωπλής τα μέσα ενημέρωσης στην ε, Δημοκρατία της Τσεχίας. Να σας υπενθυμίσω ακόμα μια φορά ότι δεν είμαστε με το ευρώ. Ε, τα μέσα ενημέρωση το αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα αρνητικά. Ακούστε κύριε Πρόεδρε. Εδώ δεν θα πρέπει να δημιουργηθούν προβλήματα και στους εμπόρους, έτσι. Εμείς έχουμε το πίν ε, και ίσως γι' αυτό πρόκειται εδώ, αυτό θα πρέπει να συζητήσουμε. Και το πρόβλημα για αυτό το θέμα δεν είναι τόσο σημαντικό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η κυρία λέει ότι θα πρέπει τα λογισμικά να προσαρμοστούν κατάλληλα και θα ήθελα να ακούσω κάτι περισσότερο για αυτό το θέμα συζήτησα με μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, και κατά γενικό τρόπο ότι εκτιμών ότι είναι ένα σύστημα που θα πρέπει να ισχύσει ιδιαίτερα γοργά και οι καταναλωτές ε, να μπορέσουν ε, εάν υπάρχουν πολλές καταθέσεις μεταφορές κλπ θα μπορούσε να πλουστευτεί το πράγμα. Ε, δυστυχώς όλες ε, οι τράπεζες το έχουν εφαρμόσει προς το παρόν και είναι πολύ εύκολο από τη στιγμή που έχετε ένα εθνικό αριθμό λογαριασμού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ακριβώς ε, και το BIC και το IBAN και η Επιτροπή στην πρότασή της αυτό υποδεικνύει ότι θα πρέπει να υπάρξει καλύτερη και περισσότερη ενημέρωση και τότε θα μπορούσε αυτή η μεταβολή να γίνει πολύ πολύ γρήγορα. Εντάξει, δεν νομίζω ότι για τον ένα ή τον άλλο καταναλωτή θα υπήρχε κάποιος κίνδυνος. Εντάξει, θα υπάρξουν ακόμα δύο ψηφία και δύο γράμματα που θα προσθεθούν και δεν αλλάζουν και πολλά πράγματα γιατί το όλο σύστημα παραμένει το αυτό. Κατά γενικό τρόπο είναι, είμαι σύμφωνο με τον κύριο Σμιτ. Θα πρέπει όσο γίνεται πιο γρήγορα να υιοθετήσουμε αυτό το σύστημα. Και επίση μεσολαβεί μακρό σύστημα προσαρμογή. Ε, το 10% συναλλαγών χρησιμοποιούν το σύστημα αυτό και θα πρέπει να υιοθετεί αυτό το γενικό σύστημα για να πάμε προς την αυτή κατεύθυνση. Δεν υπάρχει νομίζω κανονικά κανένα συγκεκριμένο πρόβλημα που να ε, αποτρέπει από την γοργή χρησιμοποίηση αυτού του συστήματος. Ο κύριος Σβάμπ, ευχαριστώ την κυρία Γκέπαρτ για την γενική της ε, εισήγηση και εμείς δεν έχουμε ακόμα συζητήσει το θέμα στην ομάδα μας. Οι συζητήσει όμω που γίνονται για τον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο πληρωμών οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι αυτή η ενοποίηση, αυτή η ενσωμάτωση των, των ευρωπαϊκών τραπεζών πρέπει να γίνει. Δεν χωράει άλλη αναβολή. Πρέπει να γίνουν αυτές οι προσαρμογές ε, σε αυτούς τους ε, πολλαψήφιους αριθμούς ε, δεν γίνεται αλλιώς καταναλωτές πρέπει να τους κατανοήσουν εάν θέλουν να εκτελούν διασυνοριακές μεταφορές χρημάτων, πληρωμές κλπ. Είμαστε υπέρ, υπέρ όλων αυτών των προτάσεων και περιμένουμε με μεγάλη χαρά τις προτάσεις κυρίας Γκέμπχαρτ. Νομίζω ο κύριος Τόν ε, έχει να σχολιάσει αυτά τα οποία ακούστηκαν. Να σας δώσω το λόγο και μετά να επιστρέψω στην κυρία Γκέπχαρτ για να κλείσουμε. Πρόεδρε, καλημέρα σε όλους. Θέλω να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο που στηρίζει αυτή την πρόταση. Όλοι παραδέχτηκαν την σημασία του να επιτευχθεί η ΣΥΠΑ αλλά δεν ξέρουν ακριβώς τι σημαίνει το να φτάσουμε εκεί. Θυμάμαι όταν ο Πίτροπος Παρνιά έκανε την ακρόασή του, εδώ και σχεδόν ένα χρόνο, είπε ότι θα υποβάλει μια πρόταση και πράγματι σβέλτα η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση και το Κοινοβούλιο έκανε δύο ψηφίσματα για να γίνει αυτή η υποβολή. Τώρα, τα θέματα που σας απασχολούν. Δύο βασικά βασικοί εμπλεκόμενοι αντιπόσκον, οι καταναλωτέ και δεύτερον οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όλο και περισσότερο ο κόσμος ταξιδεύει στην Ευρώπη για να δουλέψει, για να σπουδάσει, για να κυκλοφορήσει και χρειαζόμαστε πραγματικά ευρωπαϊκό χώρο πληρωμών. Θα διευκολύνει τη ζωή όλων μας κατά πολύ. Επίσης θα ε, αυξηθεί η αποδοτικότητα της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς. Επίσης θα υποφεληθούν πολλοί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο μικρομεσαίος τομέας στη Γερμανία είναι πασίγνωστος, αλλά η ΣΥΠΑ θα φροντίσει να βοηθήσει την απλούστευση των διαμεθοριακών πληρωμών ε, μέσω για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όλες οι βασικές ε, τραπεζικές λειτουργίες θα γίνονται από ένα βασικό λογαριασμό. Υπάρχουν πολύ μεγάλα πλεονεκτήματα όμως, όμως αν προχωρήσουμε σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σύστημα πληρωμών στην Ευρώπη, πρέπει να καταβάλουμε και ένα τίμημα. Υπάρχει ένα σύστημα δικτύου, ένα τυποποιημένο μέσο εντοπισμού των πληρωμών, αναγνώριση των πληρωμών και όπως είπε και κάποιος, η μόνη δυνατότητα είναι η χρήση του IBAN. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μην είμαστε υπερβολικοί όσον αφορά τις δυσκολίες του να προχωρήσουν προς το IBAN. Το IBAN υπάρχει σε όλα τα κράτη-μέλη και αντιστοιχεί στο υφιστάμενο ε, αριθμό λογαριασμού που μερικές φορές ε, προηγείται ο κωδικός της τράπεζας και μετά υπάρχουν δύο ε, ψηφία ελέγχου. Άρα ο αριθμός IBAN βελτιώνει και την ασφάλεια των πληρωμών και βεβαίως ε, υπάρχει και ο, ο τυποποιημένος κωδικός της χώρας, ας πούμε DE για τη Γερμανία κλπ. κλπ. Δεν είναι και τόσο δύσκολο πια. Και πολλές χώρες έχουν με επιτυχία καταφέρει να περάσουν στο ΝΑΙΠΑΝ. Το Λουξεμβούργο, η Ιταλία, το Βέλγιο κλπ. Τώρα, θα χρειαστεί χρόνο να περάσουμε στο IBAN. Και ένα από τα προβλήματα που εντόπισε η κυρία Γκέφαρτ είναι το πρόβλημα τη επικοινωνία. Υπάρχει έλλειψη επικοινωνία από το τραπεζικό χώρο, ιδίω από κάποιες τράπεζε στη Γερμανία. Και αυτό είναι ε, λυπηρό. Δεν είναι όμω πολύ αργά να διορθωθεί το πράγμα. Κάποιες τράπεζες ήδη βάζουν τον IBAN στις πιστοτικές κάρτες, κάρτες πληρωμής των καταναλωτών και έτσι είναι πολύ εύκολο να εντοπιστεί αυτό ο αριθμό το πρόβλημα είναι, είναι ότι αν υπάρχει μεγαλύτερης διάρκειας μεταβατική περίοδο, είναι διπλό. Αφενός μεν καθυστερούν τα καταναλωτικά και οικονομικά ωφέλη και από την άλλη ε, τιμωρούνται οι τράπεζες και οι χώρες που έχουν ήδη επενδύσει για να κινηθούν προς το ΣΥΜΠΑ γιατί έχουν ε, προχωρήσει. Πρέπει λοιπόν να μην τιμωρηθούν αυτοί, να κινηθούμε πιο γρήγορα. Το πρόγραμμα αυτό έχει ξεκινήσει εδώ και έξι χρόνια σχεδόν. Εδώ και πάνω από τρία χρόνια υπάρχουν τέτοιου είδους ε, πιστώσεις ΣΥΠΑ. Δεν θα πρέπει λοιπόν να πούμε ότι δεν είχε γνώσει ο τραπεζικός τομέας ότι αυτό ερχόταν. Η πρόταση της Κομισιόν είναι και ρεαλιστική και εφικτή. Δύο τελικά σημεία, κύριε Πρόεδρε, αν, δεν, μου επιτρέπετε. Το ένα, το θέμα προστασίας του καταναλωτή. Βεβαίως, η πρόταση έχει κάποιες ε, πτυχές προστασίας του καταναλωτή για να εξασφαλίζονται οι καταναλωτές όταν χρησιμοποιούν το ε, Ευρωπαϊκό Σύστημα Άμεσης ε, Χρέωσης. Δεύτερον και τελευταίο, οι, οι εταιρείε εκτός ευρώ. Βεβαίως θα θέλαμε να συμμετάσχουν στο ΣΥΠΑ όλα τα κράτη-μέλη και όλα τα κράτη-μέλη χρησιμοποιούν το ευρώ. Επειδή όμως το εθνικό ε, νόμισμα δεν είναι το ευρώ, το κόστος της μετακίνησης στο ΣΥΠΑ σε σύντομο χρονικό διάστημα είναι δυσανάλογο. Άρα για τα μη για τα κράτη-μέλη που δεν χρησιμοποιούν το ευρώ, προτείνουμε να παραταθεί ο χρόνος μετάβασης στο ΣΥΠΑ κατά δύο-τρία χρόνια. Αυτά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τις επικοδηματικές σας διευκρινήσεις οι οποίες θα μας βοηθήσουν στις λεπτομέρειες. Κυρία Γκέπαρτ, Θέλετε να ολοκληρώσετε, έχετε το χρονοδιάγραμμα ή να το κάνω εγώ. Αυτά που έχω γραμμένα είναι ότι 24 Μαΐου θα συζητήσουμε τη γνωμοδότηση. Πολύ σύντομη προθεσμία τροπολογιών 25 Μαΐου. Ψηφοφορία στην Επιτροπή 15 Ιουνίου. 27 Ιουνίου η ΕΚΟΝ θα ψηφίσει και δεν θα πάει σε καμία ολομέλεια βέβαια πριν από το Σεπτέμβριο. Θέλετε να ολοκληρώσετε. Ευχαριστώ. Να τονίσω και πάλι αυτά που είπε η Κομισιόν. Τα κράτη-μέλη εκτός Ευρωζώνης δεν αποκλείονται. Έχουν, υπάρχει μια μεταβατική προθεσμία, μια μεταβατική φάση όπου μπορούν να συμπεριληφθούν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι δεν διαιρούμε, όπως είπε ο κύριος Σμιτ, την Ευρώπη, ούτε αποκόβουμε. Ε, αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε σαφώς. Στη συζήτηση διαγρα... Ε, φάνηκε ότι υπάρχει μία διαφορά. Οι συνήθειες, ε, παραδοσιακοί τρόποι πληρωμών και οι συνήθειες που έχουμε αναπτύξει στα κράτη-μέλη είναι πάρα πολύ διαφορετικές. Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν είπε ότι μέσω της ΣΥΠΑ ή μεταφορές ε, ε, πληρωμών, μεταφορές χρημάτων υπάρχουν εδώ και χρόνια. Μα ένας Γερμανός πολίτης δεν κάνει μεταφορά, μεταφορά γραπτή, κάνει ε, μεταφορά με πιστοτική κάρτα, με τον κωδικό του. Ε, σε άλλες χώρες ε, μπορεί να γίνουν μεταφορές μέσω άλλων οργανισμών, ξέρω εγώ, ταχυδρομικών τεμιευτηρίων είναι διαφορετικά τα πράγματα και γι' αυτό υπάρχει αυτή η απόκληση. Πολύ, σημαντικά προβλήμα, πολύ σημαντικό πρόβλημα είναι η ενημέρωση των πολιτών. Ε, συμφωνώ με την Κομισιόν ότι οι τράπεζες δεν ενδιαφέρθηκαν να ενημερώσουν τους πολίτες. Αυτή τη στιγμή στη Γερμανία ε, βρισκόμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο όπου ε, το χρονικό περιθώριο είναι μηδενικό. Ε, πρέπει λοιπόν να υποχρεώσουμε τις τράπεζες να ενημερώσουν τους πελάτες τους υποχρεωτικά. Όλες οι τράπεζες πρέπει υποχρεωτικά να ενημερώσουν τους πολίτες, πελάτες, για να καταλάβουν και οι πελάτες πώς συντίθεται αυτός ο μακρύς αριθμός. Διότι οι πελάτες λένε ότι αυτά τα επινόησε η τράπεζα, μας ρίχνει ας στο κεφάλι έναν αριθμό με 25 ψηφία και μας λέει κάντε καλά. Ε, πρέπει να κατανοήσουν οι, πολίτες μας που είναι και πελάτες πώς δημιουργήθηκε αυτός ο αριθμός του ΙΜΠΑΝ. Ε, θα επεξεργαστώ λοιπόν την έκθεσή μου, θα φροντίσω να έχετε και έγκαιρα τι μεταφράσεις, γιατί όλοι αναμένουμε τη συζήτηση και εγώ θέλω να ακούσω τη γνώμη των συναδέλφων, των συναδέλφων μου. Ο πρόεδρος. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν μια πολύ, μια πολύ αρχή, καλή αρχή για αυτή τη συζήτηση. Περνάμε λοιπόν το νομοθετικό κείμενο, τροπολογία του κανονισμού για τη συνεργασία μεταξύ των ε, εθνικών αρχών που είναι υπεύθυνε για την προστασία των καταναλωτών. Η συγγήτρια για πρώτη φορά ήταν η κυρία Γκέπχαρτ. Άρα είναι κομμάτι της ιστορίας μας, της δουλειάς μας. Κυρία Γκέπχαρτ, πήρατε τώρα την ευθύνη να μελετήσετε τις αλλαγές. Έχουμε κάποιους σκιώδεις, τον κύριο Ρόσφορτ, Ποιος παίζει τώρα, είναι εδώ. Η κυρία Ρούλα. Εγώ θα καλύψω την ομάδα μου, ο κύριος Σαλβίνη. Ο κύριος Διόν θέλει να καλύψει την ομάδα του. Ο κύριος Μονιέ που είναι γνωστός και πολύ τακτικός ε, ε, θαμών της Επιτροπής μας είστε πρόσθετο. Λοιπόν, πείτε μας πώς θα προσεγγίσετε το θέμα. Σας δίνουμε το λόγο για να ξεκινήσει η συζήτηση. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι το δεύτερο σημείο που εξετάζουμε πάνω σε αυτόν τον κανονισμό για την προστασία του κανανατού, για τη συνεργασία, για ένα δίκτυο με τις δημόσιες αρχές, για την εφαρμογή ακριβώς των όσων ισχύουν στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η Επιτροπή πρότεινε μεταβολή του κανονισμού αυτού, αλλά μόνο από τεχνικής πλευράς και από νομοθετικής πλευράς, χωρίς να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής και μια, χωρίς μια κατάλληλη ενημέρωση του κανονισμού και συμφωνώ με την Επιτροπή ότι ο κανονισμός αυτός θα πρέπει να αλλάξει πολύ γρήγορα και δείχνει έτσι και το τι γίνεται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία ε, για την προστασία του καταναλωτή. Θα πρέπει να διατηρηθεί η νομοθετική εξασφάλιση σε κάθε περίπτωση και κυρίως για την οδηγία για τις ε, συμφωνίες αυτές και οι τροπολογίες της Επιτροπής για το παράρτημα του κανονισμού ε, νομίζω ότι είναι ορθές και νομίζω ότι σε αυτή τη φάση συμφωνούμε ότι χρειάζεται ένας λεπτομερέστερος έλεγχος εξέταση του κανονισμού. Γι' αυτό ακριβώς ε, προτείνω και μία ρήτρα αναθεώρησης και η Επιτροπή θα έπρεπε να, μας, ε, να συντάξει μία έκθεση εκτίμησης πριν από το τέλος του 2013 και θα πρέπει να υπάρξει ε, μία εξέταση ακριβώς επιχειρησιακή πάνω στον κανονισμό και ακριβώς στο πεδίο εφαρμογής του. Δεν νομίζω ότι η δήλωση της Επιτροπής αυτή καθ' αυτή επαρκεί. Εμείς ε, σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στη δική μας την Επιτροπή θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι θα καταβάλει ιδιαίτερε προσπάθειες στον τομέα αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης θα πρέπει να προτείνει ένα νέο νομοθετικό κείμενο ε, σχετικά με αυτό. Ταυτόχρονα με κείμενο αυτό και να έχουμε μια εξωτερική εκτίμηση που θα οργανωθεί και ταυτόχρονα ακροάσεις με όσους συμμετέχουν και να ε, παραστούμε σε αυτή τη διαδικασία πριν να έχουμε βαθύτερες αλλαγές στον κανονισμό και ένα κείμενο ακριβώς που θα βασίζεται πάνω σε μελέτες για την καλύτερη δυνατή εκτίμηση. Οπωσδήποτε το σύστημα δεν λειτουργεί τόσο καλά όσο θα έπρεπε και δυστυχώς ε, υπάρχουν κενά και συνεργασία σε πρακτικής πλευράς υπάρχουν ε, λήψεις. Πολλοί δεν συμμετείχαν καθόλου ή δεν συμμετείχαν συστηματικά, τακτικά και όπως ακριβώς χρησιμοποιούν το σύστημα, ο τρόπος αυτός δημιουργεί δυσκολίες. Οι περισσότερες από τις δυσκολίες προέρχονται από τα βασικά γιατί υπάρχουν διάφορα προβλήματα όσον αφορά τις αρμοδιότητες στην εθνική νομοθεσία για τα δικαιώματα των καταναλωτών και επειδή δεν εφαρμόζονται ομοιόμορφα υποχρεώσεις ε, δεν χρειάζεται να ε, ακολουθήσουμε τις εκκλήσεις ε, και ορισμένες πρακτικές ε, απαγορεύονται στη χώρα μέσα, όχι από εκεί προέρχονται οι υπηρεσίες Θα πρέπει να έχουμε τις κατάλληλες προτεραιότητες. Δεν μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα αποτελεσματικά εάν δεν παρακολουθούν ε, τι περιπτώσεις όπου ζητείται η βοήθειά μας. Επίσης θα πρέπει να δούμε τις κατευθυντήριες γραμμές και τις κύριες προτεραιότητες, οι διαφόρες ε, νομοθεσίες ε, ε, η, ανάλογα με τη χώρα καθιστούν δύσκολη την επιβολή κυρώσεων, υπάρχουν άλλοι που παρακολουθούν ε, από κοντά και ενώ άλλες αρχές έχουν διαδικασίες νομοθετικές, δικαστικές, ιδιαίτερα αργές, χρονοβόρες. Τώρα, εάν ε, η αρχή που ζητάει κάτι δεν μπορεί να αντέξει το κόστος, τουλάχιστον θα έπρεπε να ε, προσφύγει επί παραβάση και θα πρέπει να δούμε πώς εφαρμόζεται ο κανονισμός αντί για μικρο, μικρές αλλαγές νομοθετικές όπως προβλέπονται τώρα καλύτερα θα έπρεπε να προβλεφθεί ένα πεδίο εφαρμογής που να είναι περισσότερο εκτεταμένο, περισσότερο ευρύ και γι' αυτό ακριβώς για τους καταναλώτες η αντιμετώπιση για τα προβλήματά του. θα έπρεπε να είναι περισσότερο οριζόντια και ευρεία με περισσότερη εξέταση λεπτομεριών. Και θα πρέπει να εξεταστεί επίσης κάθε κεκτημένο λεπτομεριακά για τους καταναλωτές και ορισμένοι τομείς θα μπορούσαν να περιληφθούν, να περιληφθούν στο πεδίο εφαρμογή ε, διάφορες υπηρεσίες και νομίζω ότι υπάρχουν κενά, κενά επαναλαμβάνω σε πλαίσια τα επιχειρησιακά του όλου συστήματος και στις ρυθμίσεις και που θίγουν την αποτελεσματικότητα στο σύνολο του συστήματος. Ένα παράδειγμα. Μια προσφυγή διαρκεί πολύ μακρύ χρονικό διάστημα και αν είναι και διαμεθοριακή περίπτωση καταλαβαίνετε πολύ συχνά πρόκειται όμως για ορισμένες προθεσμίες, για ορισμένες απαιτήσει οι οποίες δεν γίνονται σεβαστές και όλα αυτά ε, σε πολλές περιπτώσεις ε, και έρευνες και δημιουργούν προβλήματα και πάντως δεν υπάρχει θετική τάση, χρειάζεται αντιστραφή αυτή η τάση να γίνει θετική και θα πρέπει να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει και θα πρέπει να παρακάμψουμε τα εμπόδια τα οποία υπάρχουν. Τα μέτρα από νομικής πλευράς είναι δεσμευτικά και θα πρέπει να διαφυλάσσουν τα δικαιώματα των Ευρωπαίων καταναλωτών. Εμείς μιλάμε τώρα εδώ για την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην ενιαία αγορά και θα πρέπει να ενισχύσουμε την ε, εμπιστοσύνη τους ε, στο πνεύμα της πράξης για, του εγγραφού για την ε, ενιαία αγορά που παρουσιάστηκε τη βδομάδα που μας πέρασε. Θα πρέπει να υπάρξει μια συνοχή στην παρουσίαση και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να καταβάλει κάθε τι προσπάθεια για να διαφυλάξει τα δικαιώματα των καταναλωτών όπως επίσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε σε αυτή την κατεύθυνση να πάει ε, παραλαμβάνω ότι έχω προτείνει ρήτρε και θα επιθυμούσατε τη, μια ρήτρα και θα επιθυμούσατε το Κοινοβούλιο να την υποστηρίξει και δεν είναι ότι θέλουμε να επιβάλλουμε σόν και καλά κυρώσει, αλλά να διαβεβαιωθούμε ότι θα διατηρηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών γιατί είναι ο ακρογωνής λήθος στο σύστημα. Ευχαριστώ πολύ. Κάναμε μια εκτεταμένη επισκόπηση του θέματος της συνεργασίας των καταναλωτών. Είναι πέρα ε, του πεδίου εφαρμογή αυτού που προτείνει η Κομισιόν, αλλά έχει σχέση με αυτό που προτείνετε εσείς οι βιολογικές σκέψεις. Θα επανέλθουμε αργότερα σε αυτό. Οπότε κάποιος από το ΕΛΚ παρίσταται. Α, κύριε ε, ναι βεβαίως. Είστε είναι επειδή κάθεστε εδώ και γι' αυτό δεν σας είδα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Την επόμενη φορά θα πρέπει να εγκατασταθώ εδώ στο κέντρο ακριβώς ε, της αίθουσας για να με βλέπετε. Εν πάση περιπτώσει, ε, θέλω καταρχήν να συγχαρώ τον εισηγητή για την ε, ολοκληρωμένη παρουσίαση αλλά και τις εξηγήσει όχι μόνο τώρα αλλά και το, την επεξηγηματική δήλωση της έκθεσης. Ο κύριος Ρίπο επεσήμανε διάφορα μειονεκτήματα στον κανονισμό CPC και άρα μια μελλοντική αναθεώρηση ίσως και να χρειαστεί υπέρ των καταναλωτών. Το θέμα είναι πότε θα γίνει. Όλοι συμφωνούμε ότι αυτό πρέπει να γίνει. Όταν φτάνουμε στην διαμεθοριακή συνεργασία, τελικά προκύπτουν πολύ σοβαρά θέματα, όπως επεσήμανε και ο κύριος Ρήπο. Παρότι ο κανονισμός CPC ήταν αναγκαίος, επειδή χρειαζόμασταν ένα εργαλείο να χειριστούμε τις παραβιάσεις ε, το, της νομοθεσίες προστασίας καταναλωτών σε διαμεθοριακό επίπεδο δεν έχει παρά τα αυτά λύσει το πρόβλημά μας. Υπάρχουν ας πούμε οι διάφοροι έμποροι απατεώνες οι οποίοι κάνουν διαμεθοριακό εμπόριο με ε, στρεβλώσεις και ε, σε βάρος των συμφερόντων των καταναλωτών. Αυτές είναι στρεβλώσεις που ο κανονισμός ο CPC κατά την άποψή μου θα πρέπει να εξαλείψει. Άρα θεωρώ ότι τα προβλήματα δεν έχουν λυθεί. Εξ όσων από την παρουσίαση που έκανε ο εισηγητής, θέλει να στείλει ξεκάθαρο πολιτικό μήνυμα, όμως χωρίς να ε, θέσει σε ομοιρία την αναθεώρηση του κανονισμού CPC για λόγους νομικής ασφάλειας. Επίσης αντιλαμβάνομαι ότι η Κομισιόν αλλά ακόμα και το Συμβούλιο επιθυμούν μια γρήγορη λύση στο ζήτημα που είναι τεχνικό και άρα η ρήτρα αναθεώρησης που προβάλλεται από τον κύριο Ρήπο είναι μια λογική ε, συμβαστική πρόταση για να κάνουμε την αναθεώρηση που θέλουμε χωρίς να χρειαστεί να γίνει τόσο ε, τώρα ε, ευκαιρία μιας τεχνικής πρότασης. Μάλλον συμφωνώ. Θεωρώ την πρόταση ε, ένα λογικό τρόπο να προχωρήσουμε. Επίσης ελπίζω ότι θα σας στηρίξει και η Κομισιόν και το Συμβούλιο. Και ελπίζω ότι μπορούν να συμφωνήσουν με την ρήτρα αναθεώρησης που μου φαίνεται λογική, να συμφωνήσουν δηλαδή μαζί μας, ώστε το θέμα να κλείσει κατά τη διάρκεια της Ουγγρικής Προεδρίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Με μεγάλη χαρά σας βλέπω στην Επιτροπή. Ο κύριος Ροσφόρ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Φτάνει να είναι στη μέση εδώ για να τον δει ο πρόεδρο. Ε, τα κεντρώα κόμματα είναι φυσική του θέση και εμεί είμαστε σαφιλέθροι σε αυτή τη θέση. Ευχαριστώ τον ε, εισηγητή που μας έκανε μια σύνοψη ιδιαίτερα πλήρη και όπω έπρεπε για το θέμα αυτό. Ναι, πρόκειται για τεχνικής φύσεως θέμα, χρειάζεται να ενημερωθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα, πάνω σε αυτό όλοι συμφωνούμε. Στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων μα είχε προτείνει ο συγητής τρεις, ε, τρία ενδεχόμενα, αλλά τα δύο από αυτά είναι σημαντικά. Πρώτα απ' όλα, ε, να υιοθετηθεί το κείμενο όσο έχει για να προχωρήσουμε όσο γίνεται γρηγορότερα. Η δεύτερη επιλογή να έχουμε πολύ λίγες ιδιαίτερα επιλεγμένες τροπολογίες, κατάλληλα και όπως πάντα σημαίνει στη ζωή όταν είναι τεχνικό κείμενο εκεί υπάρχουν ε, τροπολογίες τεχνική δεν είναι μόνο τεχνική, αλλά συνοδεύεται από ένα μένυμα με πολιτικό περιεχόμενο και κανονικό συνηθισμένο. Αυτό είναι η δουλειά των βουλευτών. Για να δούμε τώρα πώς θα καταλήγουν η μία και η άλλη στρατηγική. Εάν χωρίς καμία τροπολογία γρήγορα γρήγορα κλείσουμε το κείμενο, τότε θα ήταν, θα μας πείραζε αυτό. Γιατί τι θα σήμαινε ότι ο κανονισμός, ο οποίος απαραίτητος, απόλυτα. Είναι, καταλήγει σε μια διαδικασία ή σε δρόμους που δεν μπορούν να λειτουργήσουν κατάλληλα. Εδώ στο ξεκίνημα αυτός ο κανισμός γιατί θεσπίστηκε υπήρχαν κενά στην προστασία των καταναλωτών τα κενά δε αυτά τα είδαμε ακριβώς στον κανονισμό αυτό, έχουν να κάνουν με τη λογική διαμεθορική συνεργασία που δεν αρκεί αυτή καθ' αυτή και που θα αντικατευθεί επειδή πρέπει να υπάρχει κατάλληλη συνεργασία ανάμεσα στα δίκτυα μέσω και του κανονισμού και θα δούμε τι γίνεται. Δουλεύει καλά ή δεν δουλεύει καλά. Ναι, εντάξει, καλά τα πάει. Ε, αυτό το δίκτυο το υποστηρίζουμε πλήρω. Αλλά ίσω ε, δουλεύει λίγο λιγότερο από ό,τι θα θέλαμε σε απόλυτου αριθμού. Θα πρέπει να βελτιωθεί. Η πρώτη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το έδειχνε αυτό. Περιμένουμε και το δεύτερο τώρα που ίσως θα έχει να μας δείξει και όπως ελπίζω διάφορες βελτιώσεις. Θα πρέπει όμως ταυτόχρονα να προσπαθήσουμε ώστε να λειτουργήσει ακόμα καλύτερα. Θα αναφέρω μόνο δύο ε, οφθαλμοφανή στοιχεία. Πρώτα απ' όλα υπάρχει ανισορροπία της στατιστικής ανάλογα με το κρατός μέλος. Θα επιμείνω τώρα στο ότι εντάξει δεν θα υπήρχαν βέβαια και τέλεια κράτη που δεν θα υπήρχε καμία στρέβλωση στην προστασία των καταναλωτών ακόμη και διαμεθροί και αλλού που θα πήγαν τα πράγματα για άσχημα. Ξέρουμε ότι επειδή δεν υπάρχουν μέσα σε κράτη-μέλη, ανάλογα με κράτη-μέλη, γι' αυτό υπάρχουν τα προβλήματα. Αυτά δίκτυα και στο δεύτερο, στο οποίο επιμένω σημαντικό είναι, είναι οι προθεσμίες ε, που διαρκούν, διαρκούν πάρα πολύ. Τώρα θα πρέπει οπωσδήποτε να περάσουμε ένα μήνυμα. Θα πρέπει τα, όλα αυτά να βελτιωθούν. Το Συμβούλιο στην τελευταία ομάδα εργασία, το γνωρίζω πολύ καλά, ότι έκανε αυτή την επιλογή να υιοθετήσει το κείμενο όσο έχει. Αλλά αυτό το κάνει το Συμβούλιο γιατί είναι πιο εύκολο γι' αυτό. Και η συζήτηση που τοποθετείται πέρα από το χώρο παιδιά του Συμβουλίου και νομίζω και αυτό είναι ένα μήνυμα που προσφέρω σε όλους τους παρόντες σας και ρίπο επίσης. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, δεν θέλουμε να βάλουμε τρικλόποδια στην Επιτροπή, να τη βοηθήσουμε μέσα από αυτήν την οπτική γωνία εκεί τοποθετούμεθα. Συμφωνούμε όλοι, θα πρέπει να βοηθήσουμε την Επιτροπή να κάνει δουλειά της και ταυτόχρονα προσφέρουμε και το μήνυμα στο Συμβούλιο ότι σε μερικά κράτη-μέλη χρειάζονται, χρειάζεται μια σημαντική βοήθεια για να λειτουργήσει το ε, δίκτυο αυτό και εξορισμού επειδή είναι διαμεθοριακό. Πού παίζεται η ποιότητα στο πιο αδύναμο κρίκο της όλης αλυσίδας ε, και στα κράτη ακριβώς όπου η συμμετοχή στο δίκτυο εκεί είναι η πλέον αδύναμη, εκεί δεν λειτουργεί τόσο καλά το δίκτυο όπως θα έπρεπε να λειτουργεί. Γι' αυτό λοιπόν στηρίζω πλήρως τη στρατηγική του εισηγητή ώστε να ζητηθεί το πράγμα να λειτουργήσει καλύτερα και θα πρέπει να μπορούμε να κάνουμε και μια εκτίμηση μετά από μια ευρεία διαβούλευση όλων των ε, μέρων που συμμετέχουν και επίσης θα υποβάλω και προτάσεις ε, για διορμές αλλαγές στον εισηγητή, αλλά θα πρέπει να δούμε, να πρέπει να καταλάβει κανείς ότι ο στόχος μας είναι να βοήθουμε την Επιτροπή και δεν θέλουμε να τη στριμώξουμε ακριβώς τα σκηνιά με αυτά που προτείνουμε και με τις απαντήσεις που περιμένουμε. Και θα ολοκληρώσω λέγοντας ότι το τεχνικό αυτό κείμενο εντάσσεται στη φιλοσοφία των όσων εδώ στην Επιτροπή κάνουμε για την πράσπιση των καταναλωτών και κυρίω για την περίφημη αυτή οδηγία για αυτού, του καταναλωτέ, που πρέπει να κάνουμε τις κατάλληλε ενέργειε για να προσπαθήσουμε σε μια, στα πλαίσια μια εναρμόνιση. Όλα αυτά προς αυτήν την κατεύθυνση πηγαίνουν και ανήκουν και στην αυτή στρατηγική. Σας ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ κύριε Ρούλα. Ε, πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Υπήρχε μία παρεξήγηση σε εμά για το ποιος θα κάνει ή όχι την ε, γνωμοδότηση. Ε, τελικά εγώ θα το κάνω, τη σκιώδη δηλαδή. Και θα ήθελα να ακούσω και την άποψη της Κομισιόν, εφόσον εγώ θα το αναλάβω. Η Κομισιόν ζήτησε να συναντηθεί μαζί μας, αλλά δεν μπορούσα γιατί εγώ νόμιζα ότι η κυρία Τούλαν θα το κάνει. Ε, Τέλο πάντων έγινε αυτή η παρεξήγηση. Θα ήθελα να ξέρω τις απόψεις της Κομισιόν ε, πού θέλει την ενίσχυση τη δική μας και τι ακριβώς ζητάει. Ο Πρόεδρος, εκ μέρους της δικής μου ομάδας, ε, συμφωνώ σε πολλά με τον κύριο Μπουσοτήλ, Έχουμε τακτική ενημέρωση από τον κύριο Μόλνερ και την ομάδα του. Σίγουρα θα τονίσει ότι ε, εδώ ολοκληρώνουμε και βελτιώνουμε την υπάρχουσα νομοθεσία και καλύπτουμε ορισμένα κενά. Μπορούμε λοιπόν, πιστεύω, να προχωρήσουμε γρήγορα στο να καλύψουμε αυτά τα κοινά ε, αλλά ορισμένα ε, θέματα πρέπει να τα μελετήσουμε ειδικά εν ώψη της μελλοντικής στρατηγικής. Η δική μου άποψη είναι να προχωρήσουμε γρήγορα γιατί θα έχουμε πολλές δυνατότητες συζήτησης και βέβαια μπορούμε να συντάξουμε πάντοτε και μια πολιτική έκθεση. Πάντως πρέπει να αρχίσουμε τη δουλειά για την πολιτική των καταναλωτών είναι σημαντικό θέμα. Ο κύριος Διόντς έχει κάτι να πει. De Jong. Ευχαριστώ. Ε, δεν συμφωνώ απόλυτα, διότι επισήμως δεν έχουμε σκιώδη σε αυτή την έκθεση, γιατί έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στον εισηγητή μετά τη συζήτηση βέβαια που έγινε εδώ και έχοντας διαβάσει και τη γνωμοδότηση πιστεύω ότι έχουμε δίκαιο που δεν ε, ορίσαμε σκιώδη εισηγητή γιατί ε, συμφωνούμε με τον εισηγητή και ε, υποστηρίζουμε απόλυτα τις απόψεις του. Και τέλος η κυρία Γκέπαρτ που ήταν η πρώτη εισηγήτρια σε αυτό το θέμα. Θα είμαι σύντομη. Έχω μόνο ένα ερώτημα στην Κομισιόν, αλλά συγχαίρω και τον εισηγητή μας, τον κύριο Μήτρο Ρέπο. Το συγχαίρω για την πρότασή του, διότι μας ε, ακολουθεί ακριβώς το δρόμο που είχαμε προτείνει τότε στην τροποποίηση, στο, στον κανονισμό. Δηλαδή έναν απλουστευμένο τρόπο υλοποίησης ε, των διατάξεων αυτών στα κράτη-μέλη. Και είχαμε αντιταχθεί έντονα στο Συμβούλιο, ο οποίος ε, είχε φέρει μεγάλη αντίσταση. Ε, υπήρχαν πάρα πολύ σημαντικές διαφορετικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Έλειπε και η εμπιστοσύνη μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών και είχαμε πει ότι θα κάνουμε αυτές τις αξιολογήσεις διότι ε, από τη στιγμή που θα αρχίσουν να συνεργάζονται οι αρμόδιες αρχές και οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί και ενώσεις, θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια πιο απλουστευμένη διαδικασία. Το υπήρχε πραγματικά ε, μεγάλο γραφειοκρατικό βάρος, αλλά τότε δεν γινόταν αλλιώς. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω την Κομισιόν, πότε πιστεύετε ότι θα επιτύχουμε μία απλούστευση του κανονισμού, μία απλούστευση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών. Ε, μελετώντας την πρότασή σας βλέπω ότι δεν θα γίνει αυτό σύντομα διότι αντιμετωπίζεται ακόμα μεγάλες δυσκολίες. Μετά λοιπόν από αυτή την τροποποίηση του κανονισμού πότε πιστεύετε ότι επιτέλους αυτή η συνεργασία θα ε, απλοποιηθεί για να επωφεληθούν και οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές. Ωραία. Ο κύριος Μόλνερ. Και μετά θα ολοκληρώσει ο εισηγητής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τα μέλη της Επιτροπής. Θέλω να πω ότι είμαι ευγνώμων για όλα τα σχόλια. Ε, αισθάνομαι ότι φροντάζετε τα συμφέροντα των καταναλωτών. Θέλετε να φτιάξετε έναν καλύτερο κόσμο για τους καταναλωτές. Ο σκοπός σας είναι να βελτιώθει η κατάσταση για όλους. Το παράρτημα του κανονισμού CPC για το οποίο συζητάμε και αποτελεί τον βασικό στόχο της πρωτοβουλίας απαιτεί ενημέρωση. Η πρόταση της Κομισιόν είναι τεχνικής φύσεως αντικατοπτρίζει μόνο τις νομοθετικές ε, αποφάσεις που λήφθηκαν αλλού σε κάποια άλλη στιγμή. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι εντάξει αυτά είναι όλα και όλα τα άλλα είναι ωραία και καλά και δεν χρειάζεται τίποτα. Αλλά δεν ισχύει αυτό. Η Κομισιόν δεν ισχυρίζεται ότι όλα λειτουργούν θαυμάσια στον τομέα του CPC. Δεν θέλουμε να κρύψουμε ότι υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Επίσης πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι τα ζητήματα αυτά δεν είναι νομοθετική φύσεως κατά ανάγκη. Ας μην το ξεχνάμε αυτό. Συγκέντρωσα με προσοχή τα παραδείγματα που έδωσαν τα μέλη της Επιτροπής. Όταν μιλήσαμε για διαφορετικές προθεσμίες, πόσο χρόνο χρειάζεται η έρευνα, πρέπει να παραδεχτούμε, όπως επεσήμενε και η κυρία Γκέπχαρτ, ότι υπάρχουν πολύ διαφορετικές νομικές καταστάσεις. Σε πολλές χώρες οι έρευνες αυτές είναι ποινικέ νομικού δικαίου, οπότε πρέπει τα νομικά, τα νομικά επίπεδα να είναι πολύ ψηλά. Σε άλλες είναι διαδικαστικές διαδικασίες ή και απλουστευμένες διαδικασίες, οπότε μιλάμε για εβδομάδες ή μήνες. Τα δικαιώματα σε κάθε περίπτωση είναι πολύ διαφορετικά ανάλογα με το είδος της διαδικασίας. Οπότε είναι πράγματα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν μιλάμε για εναρμονισμένη προσέγγιση ε, στις προθεσμίες. Οι προτεραιότητες. Οι προτεραιότητες είναι πολύ σημαντικές, διότι ακριβώς σε αυτές στηρίζεται η καταναλωτική πολιτική της Ευρώπης. Θεωρώ ότι κάθε υπεύθυνη κυβέρνηση και διοίκηση θέτει τις δικές της προτεραιότητες και κάθε χρόνο γίνεται στην Επιτροπή ΣΥΠΙΣΗ μια συζήτηση. Μιλάμε με τα κρατη και αυτούς οι οποίοι εφαρμόζουν να στείλουν ένα πρόγραμμα δράσης εφαρμογής. Αυτό είναι. Συζητείτε με τα κράτη-μέλη, στηρίζεται στην εμπειρία τους και εγκρίνεται από αυτούς. Αυτή η διαδικασία αποφάσισε το θέμα της επόμενης συζήτησης. Πόσα σεμινάρια θέλουμε να οργανωθούν επίσης αποφασίζεται οι προτεραιότητες δεν είναι καινούριο στοιχείο στη CPC. Ήδη σε πρακτικό επίπεδο υφίσταται. Δεν είμαι απολύτως βέβαιος πώς μπορεί το ζήτημα να αντιμετωπιστεί με νομοθετικό τρόπο και να βελτιωθεί. Σαφώς είναι ευπρόσδεκτα αυτά που είπε ο κύριος Μπουζουτήλ, δηλαδή η πρόταση αυτή να μην γίνει όμοιρος πολιτικών διαμαχών. Δεν το θέλουμε αυτό, ούτε το Κοινοβούλιο, ούτε το Συμβούλιο, ούτε η Κομισιόν. Το ερώτημα που τίθεται είναι πώς να το λύσουμε. Όλες αυτές ε, οι βελτιώσεις που γίνονται αφορούν το νομοθετικό κείμενο ή αφορούν την εφαρμογή, τις εθνικές διαδικασίες δηλαδή, τον τρόπο με τον οποίο ε, συνεργάζονται τα κράτη-μέλη. Αν ισχύει το δεύτερο, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί το ζήτημα μέσω νομοθετικής πρότασης. Βεβαίως, πρέπει να γνωρίζουμε ότι μπορεί να υπάρξει νομοθεσία που να μην χρησιμοποιείται πολύ συχνά στο πλαίσιο του CPC. Άρα διαρωτόμαστε αν βρίσκεται σωστά ως παράρτημα του κανονισμού CPC. Υπάρχει νομοθεσία που για κάποιους λόγους έχει παραληφθεί και, δεν, και θεωρούμε ότι θα έπρεπε να είχε συμπεριληφθεί. Δυστυχώς από σήμερα δεν έχουμε στοιχεία ούτε υπέρ ούτε κατά ε, για κάποιο νομοθετικό κείμενο. Δεν έχει γίνει ούτε, στην, ούτε από την Κομισιόν, ούτε στα κράτη-μέλη, ούτε από το Κοινοβούλιο. Και άρα δεν μπορούμε να εντοπίσουμε κάτι που ήδη υπάρχει, δεν μπορούμε να υποδείξουμε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι υπάρχει έλλειψη κάτι για κάποιο συγκεκριμένο πράγμα. Οπότε η Κομισιόν αποφάσισε να ξεκινήσει μια διαδικασία, μια σειρά σεμιναρίων με ε, τη συμμετοχή και τις απόψεις αυτών οι οποίοι εφαρμόζουν τον κανονισμό, ποια είναι τα προβλήματα που πρέπει να επιληθούν. Αυτό θα γίνει φέτος. Ε, ένα από τα σεμινάρια αφορά τις προτεραιότητες, τον καθορισμό ε, προτεραιοτήτων, θέλουμε συνεργασία των κρατών μελών. Δεύτερον, πώς να συνεργαζόμαστε, πώς να προσφέρουμε καλύτερη ποιότητα συνεργασίας, αυτό αναφέρθηκε και στη συζήτηση. Επίσης υπάρχει και ο ρόλος του συντονισμού, τι μπορεί να κάνει η Κομισιόν για να διευκολύνει τον συντονισμό. Όλα αυτά είναι καθοδόν. Επιπλέον θέλουμε να κάνουμε μια εξωτερική αξιολόγηση για να καταλάβουμε ποια είναι τα καλά στοιχεία και ποια είναι τα όχι καλά στοιχεία. Στα πλαίσιο αυτό θέλει η Κομισιόν να κάνει μια εξωτερική δημόσια διαβούλευση όπου όλοι καλούνται να εκφράσουν απόψεις. Όχι μόνο τα κράτη-μέλη, όχι όσοι έχουν σχέση με τη διαδικασία, αλλά όποιος πολίτης, επιχείρηση ή οποιοδήποτε άλλος ενδιαφέρεται. Κατά πάσα πιθανότητα αυτό είναι και το πιο επικίνδυνο στοιχείο από άποψη χρόνου. Δεν μπορούμε να κρίνουμε πόσα σχόλια θα έρθουν. Το ανέφερα και προηγουμένως. Οι τελευταίες διαβουλεύσεις που γνωρίζω στη ΣΑΝΚΟ οδήγησαν σε πάνω από χίλιες απαντήσεις για τη διαφήμιση του καπνού, πάνω από 50.000 απαντήσεις. Πρέπει λοιπόν να, να ε, αξιολογήσουμε, αλλά δεν μπορούμε να πούμε πόσο χρόνο θα χρειαστεί η αξιολόγηση τέτοιου είδους σχολείων. Οπότε, Κατόπιν αυτού είναι ευπρόσδεκτο το ότι θα παραληφθούν οι προθεσμίες που θα επιβληθεί. Υπάρχει προθεσμία, η Κομισιόν το έχει δηλώσει δημόσια. Είμαστε πανευτυχείς να κάνουμε δήλωση, ήδη έχει γίνει στο Συμβούλιο. Δεσμευτήκαμε δημόσια, αλλά δεν μπορούμε να πούμε μέχρι πότε θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία το θέμα του πώς μπορεί το Κοινοβούλιο να βοηθήσει την Κομισιό να περάσει το μήνυμα αφορά μάλλον το θέμα των πόρων. Σχετίζεται με τους πόρους. Είναι θέμα προτεραιοτήτων. Οπότε θέλω να ρωτήσω την Επιτροπή, να, ζητήσω από την Επιτροπή να στείλει μήνυμα στα κράτη-μέλη να αντιμετωπιστούν με κατά προτεραιότητα τα θέματα προστασίας των καταναλωτών που αφορούν όλους τους πολίτες ε, πρέπει να κατευθυνθούν χρήματα προς αυτές τις δράσεις. Υπάρχει αυτός ο κανονισμός, αλλά υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι επηρεάζονται. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ. Λυπούμε που δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Not appear the television now, but both of them seem Τεχνικό πρόβλημα με τα μικρόφωνα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Πρέπει να σβήσετε το μικρόφωνο σας. Α, εντάξει. Και σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Σήξατε ε, σημαντικά θέματα και Ποτέ δεν χάσαμε την ευκαιρία να τονίσουμε τη σημασία της συνεργασίας στα ψηφίσματα, η ε, στους κανονισμούς τους οποίους υιοθετήσαμε. Η κυρία Γκέπαρτ ε, και ο εισηγητής θα ολοκληρώσει. 19 Απριλίου στις 12 το μεσημέρι, ε, προθεσμία τροπολογιών 4 εξέταση τροπολογιών 24 Μαΐου, 25 Μαΐου ε, ψηφοφορία της νομοδότησης και ολομέλεια τον Ιούλιο. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να περάσει στην Ολομέλεια πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Κύριε Σιγητά, έχετε κάτι να προσθέσετε. Πολύ σύντομα, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης ε, όλους για τα σχόλιά τους και για τις ερωτήσεις τους βέβαια. Χαίρομαι γιατί διαπιστώνω ότι για όλους μας είναι σαφές ότι η προστασία των καταναλωτών είναι και το κύριο, το καυτό εδώ θέμα. Για, πιστεύω στη συνεργασία και νομίζω ότι όλοι ενδιαφέρονται για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών. Θα ήθελα να τονίσω επίσης ένα γεγονός, ότι θα πρέπει να μπορέσουμε να εξακολουθήσουμε μέσα στο δρόμο αυτό και να ρωτιέμαι εάν θα επαρκούσε μία απλή δήλωση και μόνο. Πιστεύω ότι η ρήτρα αναθεώρηση θα ήταν κάτι το σημαντικότερο, το καλύτερο. Άκουσα αυτά που είπε ο εκπρόσωπος εδώ απέναντι και μπορώ να σας πω ότι μπορούμε να ελέγξουμε όλα αυτά. Το σημαντικό ποιο είναι να προχωρήσουμε και να μπορέσουμε να δώσουμε ένα μήνυμα σύμφωνα με το οποίο το Κοινοβούλιο ένθερμα υποστηρίζει αυτό το θέμα και αυτή την υπόθεση και θα υποστηρίξει τους καταναλωτές. Σας ευχαριστώ. Ωραία. Ε, ε, λυπούμε κύριε Ντεγιόγκ, αλλά μας πιέζει ο χρόνος. Ε, ίσως θα μιλήσετε σίγουρα σε κάποια άλλη ευκαιρία, γιατί είναι μια σημαντική γνωμοδότηση για την νομική επιτροπή. Ο κ. Μπάστο είναι εδώ, η κυρία Ρούλε μόλι έφυγε, ο κύριος Νέκ ήταν εδώ, θα επανέλθει. Λείπουν μερικοί σκιώδει. Όλοι πρέπει να είστε πολύ σύντομοι. Εγώ θα δώσω την προεδρία στην κυρία Κόμη σύντομα, διότι έχω μια άλλη υποχρέωση στις 12.30. Ε, είναι ε, ε, η έναρξη, η επικύρωση της ενίας πράξης, της πράξης για την ενία αγορά. Α, θα δώσω όμως πριν φύγω το λόγο στον κύριο Ντεγιόγκ για το σημείο 20. Καλύτερη νομοθεσία, επικουρικότητα και αναλογικότητα. Ευχαριστώ πρόεδρε, δεν θα ακρηγορήσω. Ε, είναι προσφυλές το θέμα αυτό και γνωστό στην Επιτροπή. Το έχουμε συζητήσει, οι πτυχές του σε διάφορες ευκαιρίες. Ε, συζήτησα και με τον ε, εισηγητή της Νομικής Επιτροπής, τον κύριο Καρίμ, δεν αντιτίθεται, ούτε έχει εκδιαμέτω αντίθετες απόψεις με αυτά τα οποία προτείνω η γνωμοδότηση της νομικής επιτοπής είναι λίγο ευρύτερη, δηλαδή εξετάζει τη διαδικασία πριν προταθεί ε, νομοθετική, πριν γίνει νομοθετική πρόταση από την Κομισιόν. Γι' αυτό δηλαδή διευρύνει το πεδίο της εξέτασης. Δεν έχω κι εγώ αντίρρηση να διευρύνω το πεδίο ε, μέσω τροπολογιών στη δική μου γνωμοδότηση. Ε, μία, ένα άλλο σημείο το οποίο τίθεται στο σχέδιο γνωμοδότησης νομικής επιτροπής είναι το εξής. Τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιεί η Κομισιόν πριν πριν παρουσιάσει τις εμπεριστατωμένες νομικές προτάσεις. Ε, πολλοί παραπονιούνται ότι το ερωτηματολόγιο μέσω διαδικτύου είναι πολύ ωραία ιδέα αλλά ε, δεν υπάρχει επαφή με την Κομισιόν και ε, δεν ξέρουμε ακριβώς τι αντίκτυπο έχει και γι' αυτό θα πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους επικοινωνίας. Επίσης, ε, το σχέδιο γνωμοδότησης περιλαμβάνει δύο καινοτομίες Η Κομισιόν γενικά πριν παρουσιάσει μία πρόταση εξετάζει τη μελέτη επιπτώσεων και την υποβάλληση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά ίσως θα μπορέσουμε και σε μετέπειτα φάση να συμπεριλάβουμε κάποια στιγμή να, να μελετήσουμε δηλαδή ποιε είναι οι επιπτώσεις σε επίπεδο επιτροπών και να ξανεπανέλθουμε στις προτάσεις αυτές από τη στιγμή που έχουν περάσει από την Επιτροπή και πριν πάνε στην Ολομέλεια, την... τις Επιτροπές του Κοινοβουλίου δηλαδή. Ένα από τα παράπονα που ακούω είναι ότι η Κομισιόν ε, τα κάνει όλα σωστά, αλλά το Κοινοβούλιο δημιουργεί προβλήματα διότι παρουσιάζει τροπολογίες που είναι πολύ περίπλοκες σε νομοθετικά ζητήματα. Επίσης, ε, αρκετές ε, επιχειρήσεις ε, ήρθαν σε μένα και μου είπαν ότι χρειαζόμαστε ορισμένα χρήματα για καινοτομικά προγράμματα. Η Κομισιόν μας είπε ότι ε, ότι ενδέχεται ότι εμπίπτουμε το θέμα μας ή το αντικείμενό μας εμπίπτει ε, σε ενισχύσεις αλλά δεν μπορούμε να βρούμε το κατάλληλο την κατάλληλη πόρτα να χτυπήσουμε. Εδώ λοιπόν πρέπει να λάβουμε επίσης υπόψη τη χρηματοδότηση, τις χρηματοδοτικές διαδικασίες και πρέπει οι διαδικασίες, ε, οι αιτήσει ε, να είναι εύκολες ε, και φιλικές προς το χρήστη, προς αυτούς που ζητούν δηλαδή τα κονδύλια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Ντεγιόγκο. Το λόγο έχουν οι σκιώδεις ηγητές για το ΕΛΚ Μπάστος. Κύριε Πρόεδρε, σας σας ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη γνωμοδότησή του γιατί ήταν ιδιαίτερα ακριβή, συγκεκριμένη όσον αφορά το περιεχόμενό της, η παρουσίασή του. Τώρα για τα σημεία που εξέτασε θα ήθελα επίση να ευχαριστήσω για την τοποθετησή του πάνω στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στην εκτίμηση των επιπτώσεων. Πιστεύω για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ότι στην έκθεση αυτή η προσπάθεια είναι να μειωθεί το κόστος το γραφειοκρατικό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και αν ε, είναι δυνατόν κάτι τέτοιο, τότε θα έχουμε τουλάχιστον 30% σε αιτήσια βάση εξοικονόμηση κόστους. Και αυτό είναι κάτι το πολύ σημαντικό και ενδεικτικό βέβαια της όλης καταστάσεως. Νομίζω ότι σαν τοποθέτηση είναι η πρέπουσα. Και μετά θα πρέπει αυτό να είναι προκαταρτικό πριν από τις νομοθετικές προτάσεις και αυτό πηγαίνει επίσης προς την σωστή κατεύθυνση. Σημείο 3 λέμε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια δοκιμή και μετά από την σχετική δοκιμή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ίσως αυτή η πρόταση να είναι κάπως υπερβολική. Τι σημαίνει αυτό, μήπως υπάρξει μια κάποια επικάλυψη των προσπαθειών, γιατί αυτή η δοκιμή θα γινόταν ήδη από την Επιτροπή ε, πριν την παρουσίαση της πρότασής της. Γι' αυτό χρειάζεται να δούμε πώς όλα αυτά δεχτούν αρνητικά σχετικά με μια δεύτερη δοκιμή. Δεύτερο τώρα, σχετικά με το in ή out, θα πρέπει να δούμε για την νομοθετική πρόταση, μια νέα πρόταση. Είναι καλό αυτό και να αποσυρθεί η παλιότερη πρόταση. Δεν ξέρουμε αν είναι πάντα καλό κάτι τέτοιο. Σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά θα πρέπει να το μελετάμε. Χρειάζεται να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να βελτιώνουμε την νομοθεσία. Και ακόμα κάτι, θα πρέπει να εξετάσουμε το ρόλο που ανατίθεται στην Επιτροπή για, την, ε, για τις επιπτώσεις ε, και το πώς επηρεάζουν την όλη κατάσταση και την, ε, όλη ανάλυση όπως προβλέπει άλλωστε και το ελεγκτικό συνέδριο. Χρειάζεται να δούμε και την πληροφόρηση των πληροφοριών που πάνε στους πολίτες, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και πιστεύω ότι λείπει μια παράγραφος από το κείμενο αυτό που να έχει σχέση με αυτή την ενημέρωση μέσω των ιστοσελίδων, των ε, συνδέσμων κλπ. Και αυτό λοιπόν θα πρέπει να μας απασχολεί για να ενημερώνουμε καλύτερα τους πολίτες μας. Ευχαριστώ, Βάλε, σοσιαλιστές. Ναι. Και εγώ θα ήθελα να δώσω συγχαρτήρια. Δεν θέλω να ασκήσω καμία κριτική. Ίσως ε, όπως και η προηγούμενη ομιλήτρια, μερικές μικροπροτάσεις για να συμπληρώσω. Έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν επικαλύψεις εργασίες. Έχουμε, υποβάλλουμε προτάσεις, έχουμε την νομική επιτροπή που τα παίρνουν αυτά για τις επιπτώσεις, όλα αυτά και τον Ιούνιο θα ψηφίσει. Θυμάμαι ότι είχαμε ακόμα μια έκθεση που κοιμάται στα συρτάρια της νομικής επιτροπής. Δεν ξέρω τι γίνεται ε, δεν ξέρω μήπως θα πρέπει, ε, αν θα πρέπει να πάμε στις ΗΠΑ για να δούμε τι κάνουν εκεί. Αλλά εδώ ίσως διευκολυθεί η δουλειά μας εάν ε, ξέραμε ότι δεν θα γνωμοδοτούσαμε πάντα από νομική επιτροπή και χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Ακόμα ένα σημείο, το σημείο 4. Νομίζω ότι υπερβάλλει κανείς όταν λέει ότι θα πρέπει να υπάρχει να ισχύει ο κανόνας one in, one out. Και έχουμε έτσι μια φιλελευθερή ιδέα στη Γερμανία, αλλά είναι ιδιαίτερα σχηματική, όπως λέει και η Μπαστος. Ίσως υπάρχουν ορισμένα πράγματα, εντάξει, σωστά, που υποστηρίζουμε, υποστηρίζουμε και την Επιτροπή να τα προσπαθήσει, αλλά δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να φέρνουν, να μας οδηγούν αυτόματα στο one in, one out η Επίτροπη υπέβαλε ήδη 2.200 προτάσεις πέρυσι για πλουστεύσεις. πέρυσι παραλαμβάνω και θα πρέπει να ξέρω κι εγώ όλα αυτά που θα τα βρω σε ποιο, σε μια ιστοσελίδα της Επιτροπής. Με ενδιαφέρει η 17η έκθεση για ε, καλύτερες, ε, καλύτερο κανονιστικό πλαίσιο που άπτεται της επικουρικότητας. Θα ήθελα λοιπόν σε επίμαχα θέματα να ξέρω πότε γίνονται μελέτες επιπτώσεων ε, παραδείγματο χάρη στο θέμα ε, των νέων λαμπτήρων το οποίο είναι τόσο επίμαχο τουλάχιστον στη Γερμανία. Τι έχει γίνει, έχει γίνει μελέτη επιπτώσεων. Ε, θα ήθελα λοιπόν να τα γνωρίζω αυτά. Το σημείο 7, ναι, στάθμιση, ισορροπία, πολύ σωστό. Σημείο 8, εξαιρετικό και λίγα σημαντικό. Όλοι το περιμένουμε αγωνία. Τα έντυπα αιτήσεων για τις ε, χρηματοδοτικές ε, διατάξεις θα ξέραμε, θα, θα, ήθελα να ξέραμε ε, ακριβώς ε, Πού, ποια είναι τα κέρια ζητήματα αναθεώρησης όλου του χρηματοδοτικού αυτού πλαισίου. Καλύτεροι κανονισμοί, έξυπνοι κανονισμοί, ε, όλοι και τα τρία νομοθετικά θεσμικά όργανα πρέπει να συμπεριληφθούν σε αυτή τη συζήτηση και όπου γίνεται και το κοινό, η κοινή γνώμη. από τους φιλελεύθερους έχει λόγο. Ευχαριστώ. Τι ωραία που ακούμε στο τέλος της ημέρας ότι είμαστε όλοι φιλελεύθεροι. Σε ευχαριστώ λοιπόν Ντένις και ε, θέλω να συμφωνήσω και εγώ με αυτά τα, τα, τις τελευταίες παρατηρήσεις που έκανα στην εισήγησή του και ιδίω με το σημαντικό ρόλο που έχουν να παίξουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να ξέρει κανείς την νομοθεσία για να γνωρίζει τι να κάνει. Καλύτερη ενημέρωση λοιπόν, καλύτερη δημοσιότητα, καλύτερη πληροφόρηση των μικρομεσαίων. Διότι 80% των μικρομεσαίων δεν ξέρουν ότι δουλεύουμε για αυτούς. Και εάν δεν ξέρουν τις προσπάθειες που, που κάνουμε εμείς να τους βοηθήσουμε, ε, ε, δεν μας υποστηρίζουν κιόλας. Πιστεύω λοιπόν ακριβώς ότι αυτή η γνωμοδότηση θα τονίσει την ανάγκη καλύτερης ενημέρωσης. Και κάτι άλλο που υποστηρίζω είναι αυτά που σχολίασε για τους ευρωβουλευτές. Είμαστε πολιτικοί και εν μέρη νομοθέτες, όλα αυτά περιπλέκονται. Ε, ωραία, καλύτερη νομοθεσία, λιγότερη με νομοθεσία, αλλά καλύτερη. Όχι ποσότητα, αλλά ποιότητα. Ιδίως για τις μικρομεσές που θέλουν να κάνουν διαμεθοριακές συναλλαγές, ε, βλέπουν ότι ορισμένες υποχρεωτικές οδηγίες ε, εφαρμόζονται σε διαφορετικό επίπεδο στο ένα κράτος μέλος και διαφορετικά στο άλλο κράτος μέλος με το οποίο συναλλάσσονται. Άρα, λοιπόν, ε, όπως το επιβεβαιώνει και ο καθηγητής κύριος Μόντι, πιστεύω ότι η έκθεση αυτή πρέπει να τονίσει ε, ότι χρειάζεται οπωσδήποτε η μείωση του αριθμού των οδηγιών ε, λόγω της επικουρικότητας και αν υπάρχει ανάγκη ρύθμιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο να εργαστούμε με κανονισμούς. Σας ευχαριστώ κύριε Μάντερς. Κανείς άλλος δεν επιθυμεί να λάβει το λόγο. και η αίθουσα αδειάζει σιγά σιγά. Ο εισηγητής ο Ντε Γιόγκ θα λάβει το λόγο, ούτε το Συμβούλιο, ούτε η Επιτροπή έχουν κάποιο εκπρόσωπο εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θεωρώ ότι όλα όσα ακούστηκαν ήταν πολύ χρήσιμα και επικοδομητικά. Πράγματι, στην παράγραφο 4 χρησιμοποιώ ε, αυτό που ακούστηκε ότι είμαστε ε, ε, γίναμε φιλελεύθεροι. Θα έχω προβλήματα βέβαια όταν γυρίσω στην πατρίδα μου. Πάση περιπτώσει, θέλω μια ένδειξη. Σε σχέση με αυτό το ένας, ένα μπαίνει, ένα βγαίνει. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Αν έχουμε άλλο κείμενο με την άποψη ότι δεν θέλουμε νέους κανόνες, εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητοι και θέλουμε να δούμε όλους τους κανόνες αν είναι απολύτως απαραίτητοι, τότε δεν θα είμαστε τόσο άκαμπτοι όσο είναι το κείμενο τώρα. Μπορούμε δηλαδή να συμβιβαστούμε από αυτό. Οι πληροφορίες. Πληροφορίες για την ομοθεσία. Έχουν βελτιωθεί τα πράγματα στην ιστοσελίδα, αλλά όπως είπε και ο κ. Βάιλερ, είναι δύσκολο να βρεθούν διάφορα πράγματα στο διαδίκτυο. Αν μπορείτε να συστήσετε κάτι που να διευκολύνει, που να εξηγήσει ε, σε αυτούς που ενδιαφέρονται τη συγκεκριμένη νομοθεσία στην ιστοσελίδα των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων, αυτό πιστεύω ότι θα αποτελέσει μεγάλο πλεονέκτημα. Σύμφωνα με αυτό. Επίσης, η ιδέα ε, κανονισμού αντί για οδηγίας πάντοτε ήμουν υπέρ και πιστεύω ότι πράγματι οι οδηγίες ερμηνεύονται διαφορετικά ενώ ο δρόμος για το μέλλον είναι οι κανονισμοί φυσικά όποτε είναι δυνατόν αυτό. Πρέπει να δούμε μια διάταξη, μια λύση που να μην είναι τελείως απόλυτη, όπως το one in, one out. Νομίζω ότι αναφέρθηκα στα περισσότερα σημεία και για τα περισσότερα σημεία είτε συμβιβασμός μπορεί να βρεθεί είτε μια προσθήκη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ντε Jong. Μπορείτε να με επιβεβαιώσετε ότι αυτές είναι οι προθεσμίες 20 Απριλίου στις 12 για την υποβολή τροπολογιών. Μετά τι έχουμε. Ψηφοφορία στην Επιτροπή 24 Μαΐου. Ψηφοφορία στην Νομική Επιτροπή 20 Ιουνίου και τελική ψηφοφορία τον Ιούλιο στην Ολομέλεια. Ναι. Συμφωνείτε. Και χαίρομαι που καταλαβαίνετε και Ιταλικά χωρίς ακουστικά. Σιγά σιγά όλοι μαθαίνουν Ιταλικά, καταλαβαίνουν. Ε, πολύ καλά. Να σε υπενθυμίσω ότι στις 3 και πάλι με τον Επίτροπο Μπαρνιέ για ανταλλαγή απόψεων με σχετικά με τις ψηφοφορίες μας και 2011-2012 τις εργασίες μας και πώς θα προχωρήσουμε με το, ε, με το θέμα αυτό.